Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Ας εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη, αλλά προηγουμένως να σας ενημερώσω ότι τα σημεία 11 και 15 αναβάλλονται. Μήπως υπάρχουν παρατηρήσεις ε, δεν βλέπω άλλε παρατηρήσει για την ημέρηση διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Ο κύριος Μάρτιν Σούλτ. Ε, κοινοποίησε στον Πρόεδρο την πρόθεσή του να παρετηθεί της βουλευτικής του, του έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από την 11η Ιανουαρίου του 2015. Δυνάμει του άρθρου 4 του εσωτερικού κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο η παρέτηση αυτή συνάδει με την πράξη της 20 Σεπτεμβρίου του 1976. Και μια δεν προβλεπόταν συνεδρίαση της Επιτροπής μας πριν την επόμενη σύνοδο της Ολομελίας που ακολούθησε την κοινοποίηση. Εγώ ως ε, εξέτασα την παρέτηση και εξακρίβωσα τη συμμόρφωσή της με την πράξη της 20 Σεπτεμβρίου του 1976. Ως εκ τούτου ενημέρωσα τον πρόεδρο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3. Δεν βλέπω αντιρρήσει ούτε για αυτό το σημείο της ανακοινώσεις και περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι τα τέλη το τέλος συνεδρίασης ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 12 η Ιανουαρίου, 24 η Ιανουαρίου και 30 η και 31 η Ιανουαρίου 2017 θα θεωρηθούν ε, ως εγκεκριμένα. Παίρναμε τώρα στην κοινή συζήτηση των σημείων 4 και 5 της σημερινής διάταξης κύρωση και προσχώρηση των κρατών μελών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο του 2010 της Διεθνούς Σύμβασης περί ευθύνης και αποζημιώσεων για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας αστικές υποθέσεις. Μια και ο υποφαινόμενος είναι ο εισηγητής για τα θέματα αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι μετά την ενδιάμεση μας έκθεση, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο, ε, στην ομάδα εργασία της συνεδρίας της 15ης Ιουλίου και θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος να η συζήτηση επί του κειμένου του σχεδίου αποφάσεων του Συμβουλίου, μια και υπάγονταν στη διαδικασία συνένεσης και όχι συναπόφασης. Και δυνάμει τη κατηγορηματική άρνηση του Συμβουλίου να ξεκινήσει διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεδομένης της ανάγκης να προωθήσουμε ένα διεθνές καθεστώς και όχι περιφερειακές λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή των αρχών περί και αποζημιώσεων για ζημίες που προκλήθηκαν από μεταφορά από πλοία επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συστήνω να συνενέσουμε στην κύρωση αυτή προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δηλαδή να κυρώσουμε το πρωτόκολλο 10, το πρωτόκολλο της ε, σύμβασης ε, του 2010 που αφορά την ευθύνη και τις αποζημιώσεις για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να, σχολιάσουν. κυρία Χίτλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Σβόμποντα κύριε Πρόεδρε, για τα δύο σχέδια συστάσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χορηγήσουμε τη συνένεσή μας στην κύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών στο πρωτόκολλο του 2010 της Διεθνούς Σύμβασης της σύμβασης δηλαδή περί ευθύνης και αποζημιώσεως ε, για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. Η διαδικασία για την ε, θέση ισχύ της σχετικής σύμβασης ήταν αρκετά αργοκίνητη και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αυτή την προσχώρηση. Η σχετική ε, σύμβαση του HNS είναι η τελευταία ε, σύμβαση για αστική ευθύνη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που δεν έχει κυρωθεί. Χρειαζόμαστε ένα διεθνές ε, καθεστώς που να διέπει την ευθύνη και τις ζημίες τις αποζημιώσεις για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών πλήν του πετρελαίου. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση με συνεχή συνύπαρξη δύο διαφορετικών καθεστώτων για την αυτιλιακή ευθύνη, που να είναι το ένα ευρωπαϊκό και το ένα διεθνές. Βέβαια είναι κρίμα που το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και σαφείς υποχρεώσεις των κρατών μελών για να προβούσε σε κύρωση και προσχώρηση της διεθνούς αυτής σύμβασης. Παρ' όλα αυτά, η απόρριψη του σχεδίου απόφαση του, Ευρωπαϊ του, Ευρωπαϊκ... του Συμβουλίου κατά πάσα πιθανότητα θα παρεμποδίσει και δεν θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και θα, μας, θα φέρει τα κράτη-μέλη σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα, ιδιαίτερα αυτά που προσχώρησαν ήδη στην ε, σύμβαση του HNS. Με την χορήγηση της συνένεσης μας λοιπόν για την κύρωση και την προσχώρηση, ίσως ασκηθεί και πίεση στα κράτη-μέλη να το πραγματοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφύγουμε το κενό που δημιουργείται από την παράλληλη συνύπαρξη δύο καθεστώτων περί και αποζημιώσεων. Αυτά. Ευχαριστώ. Μήπως το Συμβούλιο θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οπότε να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Μαρτίου φέτος. Και μια και έχουμε τη διαδικασία συνένεσης με βάση το άρθρο 99 του εσωτερικού κανονισμού, οι τροπολογίες στην Επιτροπή θα είναι παραδεκτές μόνο εφόσον στόχο έχουν την αντιστροφή της πρότασης, της σύστασης του εισηγητού. Οπότε διεκπεραιώνουμε τα σημεία 4 και 5, προχωράμε στο σημείο 6 και θα ήθελα να δώσω την Προεδρία για λίγο στον κύριο Καβαντά. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνούμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε αντίρρηση, το οποίο προβλέπει συνοπτική παρουσίαση από πλευρά μου των αποτελεσμάτων του τριμερούς διαλόγου για την φορητότητα. 7 Φεβρουαρίου καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τον κανονισμό για τη φορητότητα για την οποία μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι. Καλά νέα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί ήταν ε, ένα κείμενο που περιμέναμε, ένα κείμενο συγκεκριμένο ε, που μπορεί να επιτρέψει στον κάθε Ευρωπαίο που μετακινείται, γιατί πάει διακοπέ, γιατί ε, μετακινείται για λόγους επαγγελματικού ή ακολουθεί ένα πρόγραμμα Εράσμου. του επιτρέπει λοιπόν να έχει πάντα πρόσβαση στο διαγραμμικό περιεχόμενο της χώρας προελεύσεώς του και να το μεταφέρει αυτό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον βεβαίως έχει τη σχετική συνδρομή στη χώρα προελεύσεως και μάλιστα θα μπορεί να έχει και πρόσβαση στο περιεχόμενο του κράτους μέλους στο οποίο μεταβαίνει προσωρινά. Για να έχει μια μεταβατική ενδεχομένω διαμονή. Αυτή είναι η ουσία. Οι διαπραγματεύσεις, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή είχαν και κάποια ένταση, πρέπει να σας ενημερώσω, όχι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου όλα πήγαν αρκετά απρόσκοπτα, αλλά από πλευράς του Συμβουλίου που είναι κάπως πιο ε, διαφορετική εικόνα. Ένας ε, πρεσβευτής ε, με όλο το σεβασμό που του οφείλουμε δεν ε, μπορούσε να έχει γνώση της εντολής που είχε λάβει ε, και έτσι πολλέ φορέ χρειάστηκε να προσφύγει στην Επιτροπή αλλά και σε εμά ακόμη για να προσφέρουμε βοήθεια και πάση περιπτώσει ακόμη και με αυτό μπορέσαμε να οδηγήσουμε σε επιτυχή κατάληξη την ε, συζήτηση και το κείμενο το οποίο είναι πιστό στα όσα έχει ε, ψηφίσει η Επιτροπή μας. Συμβιβαστικές λύσεις βρέθηκαν μεταξύ των θεσμικών οργάνων, δεν σας ξεχνιάζουμε αυτό, πάντα στο Κοινοβούλιο έμεινε πιστό στην ψηφοφορία της Επιτροπής μας και έτσι οι αρχές που είχαμε ορίσει έγιναν σεβαστές. Έχουμε ένα κείμενο λοιπόν συγκεκριμένο με απτή ε, αξιοποίηση, όχι ένα αφηρημένο γενικόλογο νομικό κείμενο που δεν θα έχει καμιά εφαρμογή και γι' αυτό είμαι και ικανοποιημένο για το αποτέλεσμα. Και ευχαριστώ τους, ε, τα μέλη των διαφορών ομάδων που μας βοήθησαν. Στην ουσία τώρα. Άρθρο 1 σε κράτος μέλος διαμονής. Έχουμε εξασφαλίσει την κατάργηση της μνήας που αναφερόταν σε μια τακτική επάνωδο στην χώρα μέλους. Απλούστατα γιατί η... το Google μας παίρνει τηλέφωνο, λέει ο πρόεδρος. Για τον λόγο λοιπόν ότι δεν ε, θελήσαμε να μετατρέψουμε έναν ε, πάροχο διαγραμμικής πρόσβασης σε ελεγκτή της διαμονής ενός ε, πολίτη. Άρα καταργείται η σχετική μνήμα. Άρθρο 1 Δέλτα. Προσωρινή παρουσία σε κράτος μέλος. Εδώ δεχθήκαμε αντισταθμιστικά την μνήμα που υπενθύμιζε ότι η περίοδος της προσωρινής διαμονής πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά και αυτή τη διατύπωση διατηρούμε. Ε, δεν θα ορίσει ο νομοθέτης αν είναι δύο μήνες ή κάποια άλλη διάρκεια η προσωρινή διαμονή. Ε, θα πρέπει και ο πάροχος να ε, συμμορφωθεί βέβαια στο πνεύμα και το γράμμα του νομοθετικού κειμένου. Επίσης, για να μην αρχίσουν να πτήσονται συμβάσεις οι οποίες θα όριζαν περιορισμούς ε, συγκεκριμένους ε, της διάρκειας σε ημέρες ή μήνες, όπως έλεγα νωρίτερα, της φορητότητας, το Κοινοβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσει τη διατήρηση της εναρμόνισης που έχουμε αυτή τη στιγμή στο άρθρο 5, ε, πρόβλεψε μία παράγραφο που απαγορεύει στον πάροχο διαγραμμικής υπηρεσίας να αρνηθεί σε έναν συνδρομητή την πρόσβαση στη φορητότητα ή να την περιορίσει χρονικά. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ε, μια ad hoc απόφαση η οποία θα περιόριζε την ε, πρόσβαση στο δικαίωμα, στα δικαιώματα που προβλέπει το κείμενο αυτό, γιατί ουσιαστικά θα, τα, θα το εξετατέρωνε. Αυτό συζητήσαμε επί το πλήστον ε, άρθρο 3α μέσα επαλήθευσης της υλοποίησης με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναφέρονταν σε τρεις τρόπους, μάλιστα τόσο πολλούς που τελικά δεν μπορούν να είναι και αξιόπιστοι. Και έτσι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια απλή απόδειξη με ταχυδρομική επιστολή ή άλλη απόδειξη όπως λογαριασμό ε, ηλεκτρικού κτλ. Ε, που αποδεικνύει την διεύθυνση διαμονής του συνδρομητή. Η απόδειξη λοιπόν που επιβεβαιώνει την διεύθυνση του συνδρομητή το κράτος μέλος ή τη διεύθυνση IP Internet Protocol, η οποία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαγραμμικές υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο δεν ήθελε να υποβαθμίσει την ποιότητα των μέσων επαλήθευσης, γιατί ολόκληρο αυτό το σχέδιο έχει να κάνει με την επαλήθευση και την ε, εμπιστοσύνη, άρα προβλέπουμε σαφείς τρόπους επαλήθευσης. Στις συζητήσεις που είχαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μπορέσαμε να καταλήξουμε στην εξή ε, συμβαστική λύση, αποδεκτή. Πρώτον, ότι αυτοί οι τρεις τρόποι επαλήθευσης δεν μπορούν μόνοι τους να χρησιμοποιηθούν εάν αξιοποιούνται ως μέσα επαλήθευσης. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνεται διασταυρούμενη επαλήθευση με ένα από τα αξιόπιστα κριτήρια που προβλέπει το κείμενο και ενώ όλο αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε στον πάροχο της πρόσβασης, ώστε να επαληθεύει ότι δεν τον κοροϊδεύει ο συνδρομητής, χωρίς πάλι όμως να θέλουμε να κάνουμε μία μορφή ιωνία αστυνομική επαλήθευση ε, της ε, κινητικότητας ενός συνδρομητή ή των ε, περισσότερων της μίας διευθύνσεων που ενδεχομένω σωρεύει, με μέσα άλλωστε που δεν θα είχε ο παρόχος. Και επίσης η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3α, ίσως να το θυμάστε, πρόβλεπε αρχικά ότι στο πλαίσιο του κανονισμού η επαλήθευση από πλευρά του κράτου μέλου τη διαμονή θα μπορούσε να γίνεται κατά τη διάρκεια της ισχύω μια σύμβασης και έτσι αν έχει ε, αιτιολογημένες αμφιβολίες ένα πάροχο για την διαμονή του συνδρομητή του, θα πρέπει ο ίδιος, ο πάροχο να προβαίνει στους ελέγχους. Δεν ε, με ικανοποιούσε τόσο αυτή η προσέγγιση, γιατί η ιδέα της φορητότητας δεν μπορεί να είναι πραγματική προστομένη αξία για τον συνδρομητή παρά μόνο εάν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίζονται και γρήγορα μάλιστα οι ε, περιπτώσεις απάτης από κάποιον που θα το επιχειρούσε. Και εδώ έχουμε και την παράγραφο 4 που συζητήθηκε επί μακρόν και διαμακρόν η παράγραφος λοιπόν αυτή που, προτείναμε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή που είχε προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο. Πρόβλεπε δηλαδή τη δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων να ε, παρετηθούν από τα μέσα επαλήθευσης. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είχα υποστηρίξει την ε, γνώμη αυτή, είχα αντιταχθεί δηλαδή στη σύνταξη της σχετικής παραγράφου, γιατί οδηγούσε σε πιθανές ερμηνείες που συνιστούσαν κατά την ε, άποψή μου κίνδυνο σοβαρών παρεκτροπών στην παροχή των υπηρεσιών. Μια πλατφόρμα, παραδείγματα, η οποία θα απαιτούσε από έναν συνδρομητή αδύναμο στην ε, σύμβαση να παρετηθεί, αν δίμαναμε μέρος της σύμβασης, να παρετηθεί από το δικαιώματά του, δεν θα ήταν ε, σύμφωνοι με το πνεύμα του κανονισμού, μπορέσαμε να περάσουμε αυτή την πρόταση. Ήταν μια κόκκινη γραμμή βέβαια για το Συμβούλιο, αλλά μπορέσαμε να αντισταθούμε και έτσι να εξασφαλίσουμε την προσέγγιση των δικών μας, στις δικές μας θέσεις του Συμβουλίου, αυτό που σας ανέφερα δηλαδή, και έτσι προβλέπουμε μια νέα αιτιολογική σκέψη, την υπαριθμο 23 23C, η οποία θα περιληφθεί στο κείμενο του κανονισμού, προσδιορίζοντας το άρθρο 3 παράγραφος 4 και θα λέει ότι αυτό μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επί παραδείγματι, όταν όλοι οι δικαιούχοι των οποίων το ε, περιεχόμενο στο οποίο έχουν δικαίωμα από έναν παροχό παροχής υπηρεσιών δέχονται συνολικά όλοι να γίνεται να ε, εξαιρεθούν από την επαλήθευση από το κράτος μέλος, τότε ναι μπορεί να είναι δεκτό αυτό. Εάν ένας και μόνος αντισυμβαλόμενος μικροκαταναλωτής του ΣΥΠΗΝ αρνηθεί τότε θα ισχύει το άρθρο 3α. Δηλαδή δίνουμε και τη δυνατότητα αλλά και το μέσον ελέγχου. Ώστε κάποιος ο οποίος δεν θα έχει σοβαρά μέσα πίεση αναντι μιας επιχείρησης παροχής δραγμικών υπηρεσιών να μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και εδώ σας αναφέρω μόνο τα πιο σημαντικά ζητήματα που συζητήσαμε στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου και που έχουν συγκεκριμένη, συγκεκριμένο αντίκτυπο στην εφαρμογή του κανονισμού. Παραχωρήσεις βεβαίως και κάναμε προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αφού είναι συμβαστικό αποτέλεσμα αυτό το κείμενο. Και μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και εμείς την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε κάποιες νίκες ή μικροπαραχωρήσεις από πλευρά των του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ενώ όλο το κείμενο είναι καλό, θα κυρωθεί στην Ολομέλεια από το Σύνολο των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο, αν δεν απατώμε. Και πρέπει να πω καταλήγοντας ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανο που μπόρεσα να αναλάβω το θέμα αυτό εκ μέρου σα, εκ μέρου ε, τη Επιτροπή ΔΕ και του Συμβουλίου. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και έτσι θα έχουμε ένα καλό κανονισμό που θα είναι όλων των πολιτών που θέλουν να μετακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα συμβάλλει θετικά στην λειτουργία της Ευρώπης και την κινητικότητα πέραν των εσωτερικών σύνορων. Πολλές ώρες δουλειάς, καλό το αποτέλεσμα όμως και θα το επαληθεύσουμε με την ψήφο στην Ολομέλεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω βέβαια ότι με καταλάβατε αν υπάρχουν άλλα ζητήματα και είμαι στη θέση σα και εγώ και το επιτελείο μου. Σχόλια έχετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εσάς και τους συναδέλφους ε, που έλαβαν μέρος και συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του πολύ θετικού αποτελέσματος του τριμερούς ε, διαλόγου. Ο κύριος Νεγκρέσκος, ο σκιώδης συγκητής μας, απουσιάζει, γι' αυτό επιτρέψτε μου να διαβάσω στα αγγλικά το δικό του κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα πρώτα, τα πρώτα βήματα προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση στο επικοινωνικό περιεχόμενο δίνοντα την ευκαιρία στους Ευρωπαίους που ταξιδεύουν, έχουν δουλειέ ή σπουδάζουν, έχουν πρόσβαση σε επικοινωνικέ υπηρεσίες όπως μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίε και άλλα τέτοια προϊόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε έναν κανονισμό χωρίς χρονικό περιορισμό για όσους ε, ταξιδεύουν ε, στην Αλοδαπή με πολύ καλές ασφαλιστικές δικλείδε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και ένα κλειστό κατάλογο που περιλαμβάνει το πολύ δύο ελέγχους με, με περιορισμένη χρήση του ελέγχου της, ε, του IP, IP. Έτσι έχουμε ένα πραγματικό γνώμονα για, τη για τους χρήστες ε, επιγραμμικού περιεχομένου με, ένα... με μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία και ελπίζω να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα οι πολίτες για να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο και πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι. Εμείς σας ευχαριστούμε. Διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας και στον κύριο Νεγκρέσκου. Άλλος κανείς παρακαλώ θα ήθελε το λόγο. Ουδής. Οπότε, τι να θεωρήσω, ότι βαρεθήκατε τη φορητότητα, έχετε κουραστεί ή μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να προσθέσει κάποιο σχόλιο, παρόλο που ολοκληρώθηκαν βέβαια οι διαπραγματεύσεις. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ζήλο για το θέμα αυτό, κανείς, συμβούλιο. Ένα, αυτό είναι το όφελος του τριμερούς διαλόγου. Ε, καταφέρει να κατασβέσει όλες τις φωνές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμότατα όλους τους συναδέλφους ε, για τη βοήθειά τους. Περνάμε στο σημείο 7 και το λόγο έχει ο κύριος Ράντεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από μια εργόδη προσπάθεια και ένα χρόνο μετά την υποβολή του εγγράφου εργασίας ε, για τις ελάχιστες προδιαγραφές ε, και απαιτήσεις ελάχιστου κανόνες ό,τι αφορά το, την πολιτική δικονομία, θα ήθελα να σας παρουσιάσω επιτέλους το πιο αριστικό σχέδιο. Ε, βέβαια, ε, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτή η πρόταση. Ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με μία μελέτη για την ε, προσέγγιση των ε, διατάξεων της πολιτικής δικονομίας. Τότε ε, η έκθεση αυτή είχε τον τίτλο Μετά τη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε κάποια μέτρα, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε κοινού κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε θέματα πολιτικής δικονομίας. Πόρο απέχουμε από κάτι τέτοιο και μάλιστα έχουμε ένα είδος ε, νομοθετικού ψηφιδοτού που διαμορφώνεται από την ομολογία του ΔΕΚ, από επιμέρους διατάξεις ε, με βάση το άρθρο 114 και που ισχύουν για διεθνείς και εθνικές διαφορές, αλλά έχουμε και ένα ολόκληρο φάσμα νομοθετικών μέτρων που διέπουν την συνεργασία ε, σε θέματα πολιτικής δικονομίας, αλλά αφορούν κυρίως τις διασυνοριακές διαφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται επίσης και με την ε, εκπόνηση κανόνων ε, ποινικής δικονομίας και έχουμε και σχετική συνεργασία στα θέματα αυτά. Βέβαια, τα μέτρα αυτά δεν ισχύουν μόνο για τις διασυνοριακές διαφορές, αλλά εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις ποινικέ δίκες και διαδικασίες. Η ποινική δικονομία προβλέπει την εγγύηση θεμελιώδους ε, δικαιώματος για μια δίκαιη δίκη βάσει του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του άρθρου 6 της Διεθνούς Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, ε, οι ιδιώτες στα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους σε όλα τα κρατη και να προσφεύγουν στα δικαστήρια με την ίδια ευκολία που το κάνουν και στα δικαστήρια της πατρίδας τους. Επίσης, η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των δικαστικών οργάνων και θα εξασφαλίσουν καλύτερη προστασία των προσώπων. Έτσι θα δημιουργηθεί και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που θα ευνοήσει την εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς και θα διευκολύνει και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Κάποιοι ελάχιστοι κανόνες είναι απαραίτητοι για να ενισχύσουμε και τον ενιαίο χώρο, κοινό χώρο δικαιοσύνης που εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επαναλαμβάνω, αυτοί οι ελάχιστοι κανόνες δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα εθνικά συστήματα, ούτε ολικό και ούτε καν μερικό. Απλώς θα εξασφαλίσουν ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ω εκ τούτου θεωρώ ότι αυτοί οι ελάχιστοι κανόνες ε, θα μας επιτρέψουν και την ενημέρωση, την επικαιροποίηση κάποιων εθνικών διαδικασιών, προκειμένου να έχουμε ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών ε, και των επιχειρήσεων και πιο αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα, μια και θα είναι πιο προσιτά στους πολίτες. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους πολιτικούς μας στόχους, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εναρμόνιση, μια συστηματοποίηση και μια ισχυρότερη, εντονότερη συνεργασία που θα εξασφαλιστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Και η εισαγωγή κάποιων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βελτιώσουν την ενημέρωση για τους κανόνες και τους μηχανισμούς. Θα δώσουν μια νέα όθηση και στο διασυνοριακό εμπόδιο, χάρη στην αυξημένη εμπιστοσύνη που θα ε, υπάρχει και θα δημιουργηθεί καλύτερη εμπιστοσύνη και μεταξύ των διαφόρων δικαστικών συστημάτων, ε, μια και θα υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφάλεια δικαίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο αστικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας μια οριζόντια προσέγγιση προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιους ελάχιστους κανόνες πολιτικής δικονομίας. Η έκθεσή μου περιλαμβάνει και ένα, και ένα παράρτημα και ένα σχέδιο οδηγίας στα πλαίσια του άρθρου 81 της συνθήκης, που είναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο βήμα προόδου σε αυτή την άγουσα της εναρμόνισης των ε, διαδικασιών. Πιστεύω ότι έτσι θα καταλήξουμε σε μια πιο ισορροπημένη εφαρμογή και θεωρώ, παραλαμβάνω την πρότασή μου, ως βήμα προόδου σε αυτή την προσπάθεια σύγκλησης ε, των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών και ενδεχομένως μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και σε έναν ε, πανευρωπαϊκό κοινό κώδικα πολιτικής δικονομίας. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον για όλους, γι' αυτό και προσβλέπω στη στενή συνεργασία με τους και και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τι έχει να πει η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο από την κυρία Γουάλης για το θέμα αυτό. Και μετά τους συναδέλφους, εάν θέλουν το λόγο. Πάντως ευχαριστούμε, Ακανθόδες το έργο, με ιστορική όμως αξία. Είπατε ότι πάνω από 20 χρόνια μας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθώ στο θέμα. Λέγομαι Νοραλ Τρόσνερ. Είμαι από την μονάδα πολιτικής ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να διοργανώσω μια ανταλλαγή απόψεων για το σημαντικό αυτό ζήτημα και καλωσορίζουμε, επικροτούμε την έκθεση αυτή για την πολιτική δικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμεριζόμαστε την άποψη πως τα πολιτικά δικαιώματα είναι σημαντικά όχι μόνο σε ζητήματα ποινική αλλά και πολιτική οικονομίας. Όταν έχουμε απαξίωση των δικαιωμάτων αυτών, αυτές προκύπτουν πολλές φορέ από τι αποκλήσει που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών δικαιών των κρατών μελών ο σεβασμός των διαδικαστικών δικαιωμάτων των αντιδίκων είναι κεντρική σημασίας και από αυτόν εξαρτάται ο κοινός χώρος δικαιοσύνη της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι διάδικοι πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη σε δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό τονίστηκε από την Επιτροπή επίση στην ανακοίνωσή της με τον τίτλο Δικαιοσύνη 2020 που εστιάζει σε ζητήματα εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων, διασφαλίζοντας τα καλύτερα δικαιώματα του παιδιού σε οικογενειακές υποθέσεις. Στο σχέδιο έκθεσης, διάφορα εργαλεία πολιτικής οικονομίας περιέχουν διαδικαστικούς κανόνες. Σημαντικοί είναι οι κανονισμοί για την εξυπηρέτηση εγγράφων Εδώ αναφέρομαι σε μικρές αγωγές ή κανονισμούς περί τραπεζικών λογαριασμών, αλλά υπάρχουν και άλλοι διαδικαστικοί κανόνες που μπορούν να βρεθούν σε άλλα μέσα πολιτικής οικονομίας, όπως είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες 1 ή Βρυξέλλες 2α. Επιπρόσθετα, όπως τονίστηκε ορθά στο προσχέδιο έκθεσης, Υπάρχουν κανόνες πολιτικής δικαιοσύνης, παραδείγματο χάρη στην οδηγία περί δικαίου. Η έκθεση αναφέρει πως τα διαδικαστικά πρότυπα εξελίχθηκαν επίσης στο πλαίσιο της ερμηνείας των μέσων αυτών από το δικαστήριο για να διασφαλιστεί η κατάλληλη δικαστική προστασία των πολιτών στην Ένωση στο πλαίσιο των φυστάμενων κανόνων. Η Επιτροπή πρόσφατα ανέλαβε συγκεκριμένη δράση όσον αφορά την πολιτική δικονομία. Προβήκαμε σε μια συγκριτική νομική ανάλυση μεταξύ των κρατών μελών, αναλύοντας λεπτομερώς την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού, ταυτοποιώντας περιοχές τις οποίες ενδεχομένως απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω προχωρώντας με πιο ολιστικό τρόπο επί του παρόντος αξιολογούμε τα αποτελέσματα μιας συνολικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τις πρακτικές και τους κανόνες για να διαπιστώσουμε κατά πόσον και σε ποιο βαθμό οι αποκλήσεις των εθνικών κανόνων αποτελούν εμπόδιο για την υλοποίηση των στόχων μιας ελεύθερης κυκλοφορίας δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι επίσης παρατηρητής στο ΙΕΛΑΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάστηκε σήμερα εδώ, όπως και τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στον τομέα αυτό έως σήμερα, και του σχεδίου ELI θα αξιολογηθούν προσεκτικά από την Επιτροπή για να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό απαιτείται δράση στον τομέα αυτών. Ένα δυνατό αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής θα μπορούσε να είναι πως οριζόντια δράση, όπως προτείνεται εδώ, θα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν ο περιορισμός της δράσης σε ορισμένες πτυχές της πολιτικής δικονομίας. Παραδείγματος χάρη, η διασυνοριακή technologies needs to be explored. επίδοση δικογράφων με σεβασμό προς τα δικαιώματα των διαδίκων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως οποιαδήποτε περαιτέρω επιβολή των ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων για την πολιτική δικονομία πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό προς την ποικιλομορφία του δικαίου και των νομικών παραδόσεων των κρατών μελών και επίσης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις εξηγήσεις σας. Η κυρία Νταϊάννα Βόλης, γνωστή στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μακρών μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα της Επιτροπής μας. Και μάλιστα συντονίστρια εκ μέρους της ομάδας της. Τώρα είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου και ξεκινώ συγχαίροντας τον εισηγητή για την έκθεσή του η οποία όντως καταφέρνει πολλά προς το στόχο της διασφάλισης συγκρότησης σε αυτή την υπόθεση που είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, ένα μοσαϊκό. Και πιστεύω ότι χάρη στην, έκθεση αυτή θα έχουμε μια πολύ πιο συνεκτική προσέγγιση. Ίσως ήταν μου να εξηγήσω επό λίγο το έργο του ε, της μονάδας Α για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο πριν από μερικά χρόνια και εμπνεώμενοι από αυτό το οποίο είχε καταστεί ένα κοινό εγχείρημα μεταξύ του, Ευρωπαϊκού, του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου και του δικού μας, δηλαδή διορισμός κοινών αρχών δικονομίας, θεωρήσαμε σκόπιμο, για όλους τους λόγους που εξήγησε και ο εισηγητής, να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο, στην παραγωγή ευρωπαϊκών κανόνων πολιτικής δικονομίας. Ωστόσο, μέχρι εκεί πάει η δική μας η φιλοδοξία, δηλαδή μία μορφή κειμένου ενδοτικού δικαίου με βάση το οποίο μπορεί να εμπνευστεί ο εθνικός νομοθέτης για να προχωρήσει ένα είδος ε, οδηγού για την αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων. Όπως είπα, είναι μέχρι εκεί η φιλοδοξία μας, αλλά η λεπτομέρεια στην οποία έχουμε ε, επισέλθει ίσως ξεπερνά το πεδίο της έκθεσής σας και η δουλειά μας βεβαίως θα συνεχιστεί για ένα χρόνο ακόμη συνεργασία με ομάδες εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν τους διάφορους τομείς που ακούσατε νωρίτερα. Η πολιτική δικονομία την σύγχρονη εποχή αντιμετωπίζει προκλήσεις και λόγω των εξελίξεων της τεχνολογίας, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης ε, διασύνδεσης, στον τρόπο ζωής δηλαδή που έχουμε, τον τρόπο με τον οποίο ε, ζούμε. Και αυτά τα υπογράμμισε βέβαια και ο εισηγητής. Υπάρχουν πολλοί τομεί στους οποίους οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας τα επόμενα χρόνια ιδιαίτερα στον τομέα της επίδοσης αγράφων που ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί θα πρέπει να είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για την επίδοση, αλλά και πέραν αυτής η εικονοτηλεδιάσκεψη με ασφάλεια για τις δίκες, ε, ταυτόχρονα και επιπλέον διάφορες μορφές ADR που προχωρούν διαγραμμικά δηλαδή μορφές επίλυσης διαφορών με τη χρήση του διαδικτύου σε όρους ασφαλείας. Και βέβαια η γενική διεξαγωγή της δίκης ενώπιον του δικαστηρίου. Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε, μια, σε ένα καθήκον συνεργασίας μεταξύ των διαδίκων και του δικαστηρίου. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο για περισσότερη δουλειά, ώστε να εξασφαλίσουμε συνοχή και συγκρότηση στην υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω αν η φιλοδοξία μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ε, φιλοδοξία για έναν ευρωπαϊκό κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αλλά πάντως μπορούμε να ρίξουμε τα θεμέλια μιας τέτοιας προσπάθειας. Και πάντως μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Και πάλι ευχαριστώ τον εισηγητή για το τιτάνιο έργο του σε αυτή την υπόθεση αισθάνομαι περήφανη μπορούσα να είμαι και εγώ μέρος αυτής της δουλειάς. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Και αν κατάλαβα καλά από τις διευκρινήσεις σας, παρά την πολύ αξιόλογη έκθεση, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Άλλος κανείς παρακαλώ, κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Ράντεφ για την έκθεσή του, που είναι άρτια ε, πολύ ενδιαφέρουσα γιατί κάνει και μια ιστορική ανασκόπηση αλλά ταυτόχρονα περιγράφει ε, με πολύ ακρίβεια την παρούσα κατάσταση αλλά και τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και είναι πάντα χρήσιμο να έχουμε υπόψη ότι κάθε εθνικό δικαστήριο είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πραγματικά αποδεκτή η αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε όλα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβέ εμπιστοσύνη. Και αυτή η έννοια της αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, είναι πολύ περίπλοκη. Βέβαια, σημειώθηκε πρόοδος, για παράδειγμα, στα θέματα της κατάρτισης των δικαστών, των επαγγελματιών στον χώρο της δικαιοσύνης. Για δεκαετίες ε, ε, είδαμε πώς δημιουργήθηκαν δίκτυα, πλατφόρμες για την καλύτερη κατάρτιση και ενημέρωση, που είναι πολύ θετικά στοιχεία. Και μάλιστα ήμουν πρόσφατα σε μια διάσκεψη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και πραγματικά είναι πολύ αξιόλογη η πρόοδος. Ίσως θα πρέπει να καταστήσουμε ε, πιο δημοφιλή αυτή τη ε, δυνατότητα να γίνει μια μεγαλύτερη εκλαίκευση, ώστε να αξιοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς όλο και περισσότεροι συμπολίτε μας. Βέβαια, η αμοιβαία εμπιστοσύνη προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων σε όλα τα κρατη Και θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και να ισχύουν και κάποιες κοινέ αρχές. Και η δυσκολία έγκυται στην ανέβρεση της ισορροπίας μεταξύ των εθνικών αρμοδιοτήτων, των εθνικών παραδόσεων ε, των ε, δικαστικών συστημάτων αφενός και αφετέρου της ανάγκης ε, της ελεύθερης διακίνησης που προϋποθέτει σε περίπτωση δυσκολιών την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το δίκαιο για δίκαιη δίκη και μια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη των λοιπόν χωρών μελών. Και το μέσο για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους είναι να θεσπίσουμε με υπομονή και προσοχή κάποιους ελάχιστους κανόνες. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε γενικώ την ποιότητα της δικαιοσύνης, όχι μόνο για τις διασυνοριακές διαφορές που είναι μεν σημαντικές, αλλά ευελπιστώ ότι με αυτή την προσπάθεια θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δικαιοσύνης γενικώ. Μου άρεσε λοιπόν πάρα πολύ έκθεση. Επίσης ε, λέτε ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια διασταλτική ερμηνεία των διασυνοριακών συνεπειών. Να μην μιλούμε μόνο για διασυνοριακές διαφορές, γιατί υπάρχουν άλλες πτυχές ε, που εμπλέκονται σε αυτήν την έννοια εφόσον την υιοθετήσουμε πιο διασταλτικά. Και επίση θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις νέες τεχνολογίες, ε, να στενιστούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και για την επικοινωνία, ε, για την επίδοση, να μην χρειάζεται να μετακινηθούμε για να έχουμε δικαίωμα σε δίκαιη δίκη να μπορούμε να έχουμε τέτοια δυνατότητα, αλλά όχι κατά ανάγκη να πηγαίνουμε αυτοπροσώπως, να αξιοποιήσουμε και τα άλλα μέσα που έχουμε. Επίσης ε, και σε θέματα ανταλλαγής ε, δικογράφων ή μεταβίβαση δικογράφων και εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να αποφύγουμε τις επαχθείς ε, και πολύ διαδικασίε. διαδικασίες. Έχω και μία ερώτηση και συγχωρήστε με για την αδαιμοσύνη μου. Αφορά το άρθρο 16 δεν ξέρω ακριβώς. Στο άρθρο 16 μιλάτε για το funding. Λέτε, όταν ένας ιδιώτης τρίτος χρηματοδοτεί την ε, ε, διαδικασία αυτή, την αγωγή, ποια είναι αυτά τα όρια για αυτό του ιδιώτη τρίτου μέρους και τι γίνεται σε περίπτωση που ένας τρίτος ε, χρηματοδοτεί την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια αυτής της έννοιας. Εξηγήστε μου παρακαλώ. Επίσης, ε, μία πρόταση. Θέλουμε ε, οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και άλλου κράτους μέλους και να τηρούνται οι υποχρεώσεις διαφάνειας, ε, ενημέρωσης για τις δυνατότητες που έχει ο πολίτης, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται το δικαίωμα στη διερμηνία. Δεν και αυτό το δικαίωμα απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη δίκη. Γιατί αν πάω σε ένα δικαστήριο που δεν γνωρίζω τη γλώσσα των δικαστών, των συνηγόρων και δεν καταλαβαίνω τι ε, αναφέρεται στην ε, ακροματική διαδικασία και δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, τότε τι νόημα έχει δίκαιη δίκη. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και το δικαίωμα της διερμηνίας. Επίσης, ε, οι προθεσμίες παραγραφής. Ξέρω ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε και τις προθεσμίες της παραγραφής. Γιατί θυμάμαι τι γίνεται με τα τροχιά ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα σε άλλη χώρα μέλος. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθεσμίες παραγραφής και πότε αρχίζουν να τρέχουν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν και αυτά τα θέματα να τα εξετάσουμε με προσοχή και σύνεση, αλλά να μην τα αφήσουμε κατά μέρους. Ευχαριστώ. Θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράντεφ για να απαντήσει, αλλά προηγουμένως ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Ράντεφ, για την έκθεσή του και να πω ότι είναι σημαντικό για μας, ε, τους Ευρωπαίους πολίτες, να έχουμε πρόσβαση ε, στις ίδιες υψηλές προδιαγραφές ακόμη και για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Θα πρέπει οι πολίτες ε, να έχουν στη διάθεσή τους απλά και εύκολα μέσα, εύχριστα, για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Γιατί η ευρωπαϊκή επικράτεια είναι μεγάλη. Οπότε δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στη συζήτηση των διασυνοριακών υποθέσεων, αλλά να μιλούμε για όλε τι υποθέσεις που εκδικάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, γνωρίζουν ότι είναι απλουστευμένε οι διαδικασίες ε, στι αστικέ υποθέσει και η πολιτική δικονομία, τότε θα πηγαίνουν πολύ πιο εύκολα στα δικαστήρια. Αντίθετα, αν δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί, δεν θα προσφεύγουν εύκολα στα δικαστήρια. Επίσης, και οι πολίτες θα νιώθουν ε, πιο σίγουροι και πιο προστατευμένοι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, εφόσον μπορούν να τα απολαμβάνουν ελεύθερα σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ και τα τέλη, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι δυνατή και για πολίτες ε, με χαμηλά εισοδήματα. Να μην ε, ε, υπάρχουν διακρίσεις βάρος τους. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να είναι προσιτή προς όλους τους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και στην άποψη αυτή. Θέλουμε έναν πανευρωπαϊκό, σε κάποιο απότερο μέλλον βέβαια, κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δεν αρκούν ελάχιστοι κανόνε. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί παρακαλώ για την έκθεση του κυρίου Ράντεφ. Όχι, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μα για να ολοκληρώσει. Μην ξεχνάτε την προθεσμία για τι τροπολογίε που λήγει στι 24, 24 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ η διορία για τι για τις τροπολογίες. Και τώρα ο λόγος στον εισηγητή μας, τον κύριο Ράντεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για την υποστήριξη. Εάν ενώσουμε τις προσπαθίες μας, εάν λάβουμε υπόψη όλες τις ε, ιδέες που εκφράστηκαν εδώ και βέβαια συζητήσουμε και όλες τις πιθανές λύσεις, θα βγάλουμε πιστεύω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαίο πολίτη. Για την κυρία Ντελβό και την ερώτηση σας. Μίλησατε για το άρθρο 16. Στο άρθρο 16 έχουμε προβλέψει ένα μηχανισμό διασφάλισης. Ένας εισηγητής δηλαδή ένας ε, ασφαλιστής δηλαδή μπορεί να ε, δανειστεί σε περίπτωση ε, εισαγωγής μιας αγωγής. Προσπαθούμε λοιπόν να απλουστεύσουμε αυτή τη διαδικασία προασπιζόμενη τα συμφέροντα όλων των διαδίκων και γι' αυτό αυτό που προτείνατε πιστεύω θα βρει θέση στην έκθεσή μου. Απλώς θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υλοποιήσουμε την πρότασή σας. Ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη που εκφράσατε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Παράταση για την κατάθεση τροπολογιών. 24 Μαρτίου, μάλλον όχι παράταση, εκπνοή για την κατάθεση τροπολογιών, 24 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο λάβει το λόγο να μας παρουσιάσει τη δική του πρόταση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση της Ευρωπαϊκή επιτροπή για το 2015 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έχει θεσπιστεί με βάση το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρώπων δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 2 της Συντηρητικής Συνθήκης. Και ως εκ τούτου η προσεκτική επιτήρηση των πράξεων ή παραλήψεων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν έχει ύψιστη σημασία. Στην έκθεση αυτή εμείς ε, θα ήθελα να πω ότι επιφανειακά μόνο ασχολούμαστε με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό διαπιστώνω εγώ στην έκθεσή μου, ότι επιφανειακά μόνο, γιατί κατά τα άλλα υπάρχουν παραβιάσεις θεμελιωδών ε, ε, αρχών του δικαίου και αξιών που μπορεί να επηρεάζουν και τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχείρηματο για ολοκλήρωση και πάνω απ' όλα τι ζωέ πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Στην έκθεση λοιπόν αναφέρουμε τους τομείς ε, στους οποίους διαπιστώνονται παραβιάσεις ε, της μεταφοράς σε εθνικό δίκαιο, στους τομείς της κινητικότητας των μεταφορών του περιβάλλοντος. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει 3.450 ε, καταγγελίες παραβιάσεων, πιθανών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν την Ιταλία, την Ισπανία και την Γερμανία κατά κύριο λόγο, χώρες δηλαδή για τις οποίες έχουν καταγγελθεί προς παραβιάσεις. Πρέπει να αναφέρουμε ότι από το 2011 για πρώτη φορά ο αριθμός των νέων καταγγελιών για, ε, που ισχυρίζονται ε, παραβίαση έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 9% συγκρινόμενη νόσου με, με τα νούμερα του 2014. Έχουμε λοιπόν οργανώσεις εμπλεκομένων πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων, με βάση τις οποίες εξετάζουμε αν τηρούν τα κράτη-μέλη το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αύξηση κατά 27% στον αριθμό των νέων ευρωπαϊκών πιλωτικών φακέλων που ξεκινούν το 2015. Είναι επίσης αξιόλογη αύξηση. Ο μέσος ε, όρος επίλυσης αυτών των ζητημάτων παραμένει σταθερός στο 75%. Αναγνωρίζετε βεβαίως ότι κύρια ευθύνη για την ε, πιστή εφαρμογή και υλοποίηση του ευρωπαϊκού, κράτους, του ευρωπαϊκού δικαίου ανήκει στα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απαλλάσσονται τη υποχρέωση και του καθηκοντό του για το σεβασμό του πρωτογένου ευρωπαϊκού δικαίου κατά την εκπόνηση και ε, έκδοση παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην τήρηση ημί των όρων τη λιτότητας σε σχέση με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φερρυπίν, η ιδιωτικοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων ε, για κράτη-μέλη που είναι υπερχρεωμένα, όταν επιβάλλονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορεί να συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου και διατάξεων που έχουν να κάνουν, παραδείγματι, με το άρθρο 345 τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του οποίου οι συνθήκες δεν μπορούν επουδενή να τροποποιήσουν τους κανόνες που αφορούν ε, το καθεστώς το ιδιοκτησιακό των κρατών μελών. Κάτι το οποίο προβλεπόταν ήδη στη διακήρυξη Σούμαν. Και έκτοτε περιλαμβάνεται σε όλες τις συνθήκες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνει ότι γίνονται σεβαστές οι επιλογές των κρατών μελών ως προς την κυριότητα, το καθώς κυριότητας των υπηρεσιών που παρέχουν δημόσιο αγαθό στο κοινό στους Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι εάν τα κράτη-μέλη υποχρεώθηκαν σε κάποια περίπτωση από τη λεγόμενη Τρόικα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, Διεθνές Οσματικό Ταμείο δηλαδή, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία παραβιάζουν τις ε, συνταγματικές και διεθνείς τους υποχρεώσεις προς το σεβασμό των θεμελιωδών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι κατ' ουσίαν αδύνατον να προσβληθούν αυτές οι παραβιάσεις με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές ταυτόχρονες μελέτες και σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις, καταρχάς στο πεδίο των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περιθαλψή, την ιδιοκτησία οι εξωτερικά δικαιώματα. Επίση, περιορίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, η ελευθερία τη ενημέρωση, το δικαίωμα στην κοινωνική προόνοια, το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό, τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η αρχή τη ισότητα και το κράτο δικαίου. Η Ελλάδα είναι ένα σαφέ παράδειγμα αυτή τη κατάσταση. Λόγω των μέτρων αυτών, σημαντικό τμήμα των Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή έχει ακατάλληλη, ανεπαρκή πρόσβαση στην ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παιδική φτώχεια. 37,8% των παιδιών, 37,8% των παιδιών της Ελλάδας είναι ε, σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού του 2015, συγκρινόμενο με 28,7% του 2010. Επιπλέον, ύστερα από το 2010, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση σε ποσοστά αυτοκτονιών 35% περίπου. Συγκρινόμενο με την περίοδο μεταξύ 2003-2010. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι θάνατοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τις γεννήσεις από το 2011 και με επιτυχημένους ρυθμούς. 500.000 Έλληνες έχουν αποδημήσει στο εξωτερικό για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους εργαζόμενοι. Τέτοια μέτρα, όπως αυτά που επιβάλλονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έχουν πολλές φορές ε, σαν αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό του, της διοικητικής και δικαστικής μηχανής και της δυνατότητας για υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου από πλευράς αυτών. Θα πρέπει επιπλέον να υπογραμμιστεί ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει το χαμηλό επίπεδο υλοποίησης και μεταφοράς σε εθνικό δίκαιο των προδιαγραφών και προτύπων για το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματι, οι διατάξεις για, ε, της οδηγίας για την υποδοχή 2013-2023 από ορισμένα το ίδιο ισχύει και για τους μηχανισμούς επανεγκατάστασης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης του προσφυγικού από τα κράτη-μέλη. 5% μόνο των συμπεφωνημένων στόχων για επανεγκατάσταση έχει, έχει μέχρι τώρα υλοποιηθεί. Ω εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ιδιαίτερα να επαγρυνήσει ω προ την ε, ορθή υλοποίηση των μέτρων ε, στον ε, χώρο του ασύλου και τη μετανάστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσει στις αναγκαίες διαδικασίες επί Καταλήγοντα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν τα καθήκοντά του για σεβασμό κάθε πτυχή του ευρωπαϊκού δικαίου, ιδιαίτερω όταν, ε, παράγουν, όταν ε, νομοθετούν σε παράγωγο δίκαιο ε, ή εισάγουν ε, συμφωνίες διεθνείς ή διακυβερνητικές εκτός του πεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως με το Διεθνές Νοσματικό Ταμείο επί παραδείγματι. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν επιπλέον, να αναλάβουν τα καθήκοντά τους ε, για να προσφέρουν την υποστήριξη και αρρωγή τους προς τα κράτη-μέλη, προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε περιόδους λιτότητας και δημοσιονομικών ε, περιορισμών και βέβαια με δεδομένη την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών Μάρτιος, 8 Μαρτίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας τον Απριλίο, 11 Απριλίου ή 12. Ευχαριστώ. Merci beaucoup ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Χρυσόγωνα. Η κυρία Κάφμαν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρίως τον εισηγητή κύριο Χρυσογόνου Πιστεύω πως πρόκειται για ένα γενικά καλό σχέδιο έκθεσης που αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω εργασία. Με εκπλήσει κάθε φορά εκ νέου πόσες καταγγελίες μη εφαρμογής ενωσιακού δικαίου υπάρχουν 3.450 σε ένα χρόνο. Είναι ένα σημαντικός αριθμός και πιστεύω πως πρέπει να σκεφτούμε γιατί οι τομείς της κινητικότητας των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος πλήττονται από αυτό. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να έχει αίτια, γιατί ειδικά αυτοί οι τομείς φύγονται. Φυσικά και τα κράτη-μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την κανονική εφαρμογή και μεταφορά του ενωσιακού δικαίου και πρέπει να ανταπεξέλθουν στην ευθύνη αυτή. Αλλά πιστεύω πως και εμείς ως ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να στοχαστούμε εκ νέου τι θα μπορούσε να γίνει συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο ή και ποια είναι τα προβλήματα. Θα ήθελα να θίξω ένα ερώτημα που με απασχολεί. Επειδή κάθε χρόνο εκπονούμε μια τέτοια έκθεση ως κοινοβούλιο και θα με ενδιέφερε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται έχει καταρτήσει μια επακόλουθη έκθεση στη δικιά μας έκθεση του 2014 επειδή αν εμείς ελέγχουμε την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου τότε έχουμε κάποια ανάδραση, κάποιες συνέπειες από την έκθεση που εκπονούμε. Για μένα αυτό θα ήταν ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να λυθεί επίσης υπόψη για την έκθεση του 2015. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς. Ε, θα προσπαθήσουμε να ε, λάβουμε απάντηση στις απορίες σας, κυρία Κάουφμαν. δώσω το λόγο στον κύριο Μπούντα, μετά στην κυρία που είναι πίσω από τον κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόγωνα για την έκθεσή του. Η έκθεση αυτή πραγματικά μας παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου οδηγεί σε βελτίωση των επενδύσεων και σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο στις εθνικές τους ένομες τάξεις. Πριν από λίγο συζητήσαμε για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και είπαμε ότι θα πρέπει να προβλέπει ε, παντού τι ίδιε προδιαγραφές. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την ενωσιακή νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάση και επιβόλης κυρώσεων που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μειωθεί. Αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μια τεχνική υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται πιο τακτικά ενταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των κρατών μέλων. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό μερικές χώρες να έχουν ε, νομοθεσία για συγκεκριμένα θέματα και άλλες χώρες να έχουν τελείως διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ίδια θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να εντοπίσει τα αίτια αυτής της κατάστασης. Για παράδειγμα, για το περιβάλλον. Έχουμε πρόβλημα στη Ρουμανία γιατί δεν μπορούμε να τηρήσουμε τους όρους που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν και λογικοί. Καλή έκθεση. Θα κατατεθούν φυσικά πολλές τροπολογίες, γιατί πρέπει να διορθώσουμε κάποια σημεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γνωρίζετε τη γνώμη μου για το στόχο της ετήσιας αυτής έκθεσης που ακολουθεί τους ίδιους ε, γνώμονες με τις προηγούμενες, με μικρές διαφορές, ανάλογα το πόσο φιλελεύθερος είναι ο εκάστοτε εισηγητής. Χαιρετίζω τη μνήα ε, των συνεπειών των μέτρων λιτότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια κράτη-μέλη. Βέβαια, είμαι κατά της μνήας που αφορά την ανεπαρκή εφαρμογή των κρατών μετών, των μελών του μηχανισμού της ε, μετεγκατάστασης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το μέτρο αυτό το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους λαούς χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση. Το ίδιο ισχύει, ισχύει και για τη μνήμα του χαμηλού βαθμού μεταφοράς ε, και εφαρμογή ε, των διατάξεων για τα θέματα του ασύλου. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει το ρόλο του πυρομανή πυροσβέστη. Δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα αυτά. Και θα ήταν ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει επιτέλους μια αντικειμενική έκθεση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τις συνέπειες που έχουν τα μέτρα της στην, ασφα... στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Μπορώ να σας δώσω εγώ τα αποτελέσματα. Μαζική ανεργία, ύφεση, απώλεια ανταγωνιστικότητας και όλο και περισσότερο το ανταγωνισμό από τις αλλοδαπές εταιρείες. Αυτές είναι οι συνέπειες των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τρέσκα, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ο κύριο. Α, συγγνώμη, ο κύριο, ο κύριο Τρέσκοτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές, όλα αυτά τα σχόλια που κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση κατόπιν της δέσμευσης, της αφοσίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αφοσίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της εφαρμογής όλου του εύρους του ενωσιακή της ενωσιακής νομοθεσίας η 33η ετήσια έκθεση σχετικά με, την, με τον έλεγχο της εφαρμογής του ενωσιακού νόμου δικαίου τονίζει την πολιτική επιβολή στο 2015. Ο υψηλός αριθμός παραβάσεων που παρατηρήσαμε το 2015 δείχνει πως η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή, εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στα κράτη-μέλη παραμένει μια σοβαρή πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινή διαδικασίες επί σε καταστάσεις στις οποίες τα κράτη-μέλη αποτυγχάνουν να μεταφέρουν οδηγίες εντός μιας προδιαγραμμένης προθεσμίας στο εσωτερικό τους δίκαιο ή εάν κράτη-μέλη αποτυγχάνουν να θεσπίσουν νομοθεσία ευθυγραμμισμένη με το ενωσιακό δίκαιο. Η μια άλλη κατάσταση προκύπτει εάν ένα κράτος μέλος αποτυχεί να εφαρμόσει ορθά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως βλέπουμε, οι αριθμοί είναι υψηλοί, αν και είναι αρκετά χαμηλότεροι από ό,τι σε προηγούμενα έτη. Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος τομέας ανησυχίας ήταν αυτός των διαδικασιών επί παραβάση. Το 2015 οι τομείς που πλήγηκαν παραπάνω ήταν όντως η κινητικότητα, το περιβάλλον και οι μεταφορές. Το σοβαρό πρόβλημα που, επι, που εμένει είναι η μεταφορά των οδηγιών. Η αδυναμία, η αποτυχία της μεταφοράς οδηγιών στο εσωτερικό ένομο στην εσωτερική ένωμη τάξη των κρατών μελών εντός μιας προθεσμίες ε, αποτρέποντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να αποφεληθούν από τα ωφέλη και να αποφύγουν τα μειονεκτήματα από τα οποία τους προστατεύει το ενωσιακό δίκαιο. Παρατηρώντας τον αριθμό των νέων διαδικασιών επί παραβάση το 2015 υποχώρησε ελαφρά σε σχέση με το 2014 αλλά το πρόβλημα εμένει. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει δραστική χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει πρώτα απ' όλα μέσω της καλύτερης παροχής υποστήριξης στα κράτη-μέλη κατά την μεταφορά όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει έγγραφα και σχέδια εφαρμογής και μια σειρά συναντήσεων για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την περίοδο μεταφοράς. Μετά από αυτό το στάδιο, όταν τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να αποτυχάνουν να μεταφέρουν οδηγίε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αυστηρά τον μηχανισμό που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα που είναι η προσφυγή στο δικαστήριο με αίτημα επιβολής κυρώσεων σε κράτη-μέλη. Φέτος αναφέρουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφηκε σε τρεις περιπτώσεις στο δικαστήριο ζητώντας την επιβολή κυρώσεων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το, γιατί το περιβάλλον, η κινητικότητα και οι μεταφορές παραμένουν ο τομέας με τις περισσότερες καταγγελίες και ανησυχίες όσον αφορά την μεταφορά. Θα παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτηση αργότερα τις αιτίες, αλλά μία αιτία σχετίζεται με το κόστος που υπάρχει στον τομέα αυτό, το οποίο απαιτείται για την δημιουργία υποδομών όσον αφορά την αναφορά για την έκθεση του 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στο ψήφισμα καθώς θεώρησε πως ήδη προέβησε βήματα στο παρελθόν επειδή το ψήφισμα με αναφορά στην έκθεση του 2014 και στα ζητήματα που τέθηκαν εκεί υπήρξε αντικείμενο μεταχείριση σε προηγούμενες εκθέσεις. Γι' αυτό και δεν υπήρξε η ανάγκη εκπόνηση μιας νέας έκθεση. Αυτά είναι όλα από πλευρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Μήπως ο εισηγητής θα ήθελε και πάλι το λόγο. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που λύγει στις 8 Μαρτίου. Οπότε περάμε στο σημείο 9, την εξέταση των τροπολογιών για το θέμα της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων. Το λόγο έχει η κυρία Μπερζερόν, η συγγετριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για την έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά την τύχη των ευάλωτων ατόμων στην Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, στόχο έχει να διευκολύνει την αναγνώριση των μέτρων προστασίας, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να δώσει κάποιους ε, γενικώ αναγνωρισμένους ε, τεχνικούς μηχανισμούς προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των ευάλωτων ατόμων και τους ε, ενδιαφερόμενου πανεβαίνοντες ή τους θεσμούς. Δεν προβαίνει σε ριζική μεταρρύθμιση των εθνικών νομοθεσιών. Από ανάγνωση των τροπολογιών διαπιστώνω μια μεγάλη σύμπνοια σε ό,τι αφορά την ανάγκη κοινή δράση. Και με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά εξέτασα το μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Διευκρινίζω ότι συμφωνώ με την πλειοψηφία των τροπολογιών και ελπίζω να καλυφθούν οι περισσότερες από συμβαστικές τροπολογίες που θα εκπονήσουμε από κοινού. Ε, διαπιστώνω ότι σε επιφυλάξει και του αδιασμού τη κυρία Κομοντίνη Κάτσα. Λυπούμε που απουσιάζει, γιατί μα είχε ζητήσει διευκρινήσει. Στην ε, τροπολογία 86 ζητά πρόθεση, ε, πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι γενικά και όριστα, χωρί να λέει τι είδου πρόταση ζητά, οδηγία ή κανονισμό. Και αυτή η διευκρίνηση είναι σημαντική, γιατί το θέμα αυτό καλύπτεται από την Σύμβαση της Χάγης, το Διεθνές ε, Ιδιωτικό Δίκαιο. Επίσης είχαμε πρόβλημα με την κύρωση της ε, σύμβασης αυτής. Έχει μείνει σε εμβριακή φάση. Και αν ε, ε, δεν ε, προκρίνουμε ένα κανονισμό, ε, παρόμοιο πρόβλημα θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή θα έχουμε μια οδηγία που θα εφαρμόζεται μόνο μερικώ, κατακαιρματισμένο, οπότε τι θα έχουμε ένα επιπλέον κίνδυνο, ένα, μια επιπλέον οδηγία που δεν θα εξυπηρετεί ούτε τους ευάλωτους ενήλικες, ούτε τους θεσμούς που εμπλέκονται στην κατάσταση αυτή επίσης. Ε, η συγκεκριτρία δεν είναι υπέρ τη παρέμβαση που λέει ότι θα αποδυναμώσει τη σύμβαση τη Χάγη. Ένα όμω ευρωπαϊκό κανονισμό που σε μεγάλο βαθμό θα παραπέμπει, θα εστερνίζεται τη σύμβαση τη Χάγη, ουσιαστικά την ενισχύει. Η αναζήτηση κοινών κανόνων είναι σημαντική. Οπότε νομίζω ότι μόνο με ένα κανονισμό θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Ο κανονισμό είναι το απαραίτητο νομικό εργαλείο. Σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ δράσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ε, πολύ επιφυλακτική σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία για τους ευάλωτους ενήλικες. Πιστεύω ακριβώς ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατρανώσει τη βούλησή του για σημείωση προόδου στο θέμα αυτό. Επίσης διαπίστωσα ότι η κυρία Κομοντίνη ήταν κατά της πλήρους αναγνώρισης των μέτρων προστασίας που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος. Πρόκειται για τις τροπολογίες 41, 50 και 98. Κι όμως αυτό είναι ο στόχος ε, της έκθεσης πρωτοβουλίας Δηλαδή, ε, δεν θα πρέπει με κάθε αλλαγή χώρα να πρέπει κανείς να ξαναποδείξει την ταυτότητά του. Σε ό,τι αφορά την εντολή ανικανότητα, ε, η κυρία Κομοντίνη δεν θέλει να επισημοποιείται αυτή η επιλογή της ζωής και μόνο σε κράτη που το αναγνωρίζουν θέλει να εφαρμόζεται. Πρόκειται για τις ε, τροπολογίε 100 και 103. Δηλαδή, κάποιο που έχει ε, συντάξει τη, διαθήκη του στη Γαλλία και αποβιώνει στη Μάλτα, ε, σαν να μην ισχύει η διαθήκη του πια στη Μάλτα. Ε, γιατί η εντολή της ανικανότητας είναι ένα γεγονός, είναι ένα είδος διαθήκης. Οπότε κάποιος που έχοντας ο σώστας φρένας έχει εκφράσει την βούλησή του, τη θέλησή του, θα πρέπει αυτή η θέληση να αναγνωρίζεται και σε άλλες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, συνέπειες οικονομικές και άλλες, ε, της αναγνώρισης ενός μέτρου προστασίας που ε, αναγνωρίζεται σε ένα κράτος και πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο. Η κυρία Κομοντίνη θεωρεί ότι τα έξοδα θα πρέπει να τα αναλάβει το κράτος το οποίο έχει δεχτεί την, το αίτημα. Εμείς προτείνουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας και επιμερισμού των δαπανών, γιατί είναι προφανές ότι οι φτωχότερε χώρε δεν θα πρέπει να αναλάβουν μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, να στεγάσουν και να περιθάλψουν ευάλωτου ενήλικε που είναι κάτοικοι άλλη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια χρηματοοικονομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να αποφύγουμε άδικε επιβαρύνσει. Δεν μπορώ να μιλήσω απευθεία ε, στην κυρία Μοκομοντίνη. Δυστυχώ γιατί απουσιάζει. Άλλοι συνάδελφοι ε, στι τροπολογίε 43 μιλά για τον κίνδυνο παρέμβαση με ένα νέο έντυπο εντολή ανικανότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το έντυπο είναι ένα είναι διοικητικό και αναγνωρίζει μια κατάσταση, όπως η καταγραφή μιας διαθήκης. Στόχο έχει να διευκολύνει για όλους ε, την ε, έκφραση της θέλησης ενός ατόμου. Και σας ε, διευκρινίζω ότι μόνο οι χώρες που προβλέπουν τέτοια έντολη ανικανότητας εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία του ενιαίου εντύπου που προβλέπει την αναγνώριση αυτή της έντολης και έχουμε ουσιαστικά διακριτική συνεργασία εδώ, υποσταλτική ε, ερμηνεία μάλιστα. Κάποιοι ε, προβληματίστηκαν για την ε, διάδοση κάποιων στοιχείων που αφορούν την προσωπική κατάσταση κάποιου ή την παράβαση του ιατρικού απορρίτου ή ιδιωτικών πληροφοριών. Μα με τον πιτρό που προτείνουμε απλώς ε, στο μητρό αυτό καταγράφεται ότι κάποιος ε, δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν αναφέρεται τίποτα για το ιατρικό του ιστορικό, για την, ε, ε για την περιουσία του ή καμία άλλη πληροφορία για την ιδιωτική του ζωή. Επίσης, είστε κατά του κανονισμού, αλλά δεν νομίζω να βοηθήσετε κανένα. Μήπως θέλετε ε, να γίνει η Γαλλία ένα μικρό χωριό της Γαλλικίας του Αστερίξ και να μην έχει κανέναν γύρο. Επίσης, τροπολογίες 21, 61, 67 και 83. Διαφωνώ. Δυστυχώ ο κύριο Μπούντα έφυγε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμότατα για τι τροπολογίε του και μπορώ να συμφωνήσω σχεδόν με όλε τι τροπολογίε γιατί είναι τεχνικού χαρακτήρα και διευκρινίζουν τη δική μου πρόταση. Και διαρωτώ μήπως είναι συμβολογράφος ε, ή ήταν συμβολογράφος ο κύριος Μπούντα, γιατί πραγματικά ήταν ακριβέστατες οι προτάσεις του και σαφέστατες. Ο κύριος Τζαμπάσκι, Ναγκρέσκου, Χρυσόγονος και άλλοι κατέθεσαν τροπολογίες για να διευκολύνουν ε, τη ζωή των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας. Κύριε ε, γράψω και κύριε Χρυσόγονε, συμφωνώ με, το, με την δική σας αντίληψη για το τι εστί ευάλωτος ενήλικος και συμφωνώ με την ιδέα που έχετε για τον ευάλωτο. Θεωρώ ότι ο ορισμός της σύμβαση της Χάγης είναι πολύ περιοριστικός. Θέλουμε όμως έναν ε, ελάχιστο ορισμό, αν θέλουμε πραγματικά το κείμενό μας να, να τελεσφορήσει. Γι' αυτό και συστηματικά παραπέμπω στη Σύμβαση της Χάγης σε πολλά σημεία. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Σύμβαση της Χάγης είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο ε, διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και πραγματικά κρίμα που δεν έχει κυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη. Και τώρα, θεωρώ ότι είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερψηφίσει την έκθεση πρωτοβουλία. Μπορεί να φαίνεται πρόωρη για πολλού, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει πολύ επίκαιρη δεδομένη τη ε, Εξέλιξη ε, στις κοινωνίε μας. Και νομίζω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να είναι και οραματιστής και να προβλέπει το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Ευχαριστήσαμε τον συγκητή για την πληρέστατη έκθεση, έκθεση η οποία συμπληρώνει χωρίς να αντικαθιστά τη σύμβαση. Η Επιτροπή συμμερίζεται τους γενικούς στόχους διευκόλυνσης της διασυνοριακής προστασίας ευάλωτων ενηλίκων στην Ευρώπη. Βέβαια, προτεραιότητα της Επιτροπής, πριν από οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, παραμένει η κύρωση της συμφωνίας, της σύμβασης από τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν θα ήταν πρέπει να καταθέσουμε νομοθετική πρόταση για ε, συμπλήρωση της σύμβασης όταν έχουν προχωρήσει μόνο λίγες κυρώσεις από κράτη-μέλη. Πάντως έχουμε και θετικά νέα. Τρία κράτη-μέλη τουλάχιστον πρόκειται να κυρώσουν μέσα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους τη σύμβαση το Βέλγιο μόλις πριν από μερικές μέρες την υπέγραψε και ξεκινά διαδικασίες για κύρωση. Άρα προχωρούν τα πράγματα, υπάρχει εξέλιξη και στο στάδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά να προχωρήσει σε ειδική δράση ε, στοχεύουσα στην ε, διευκόλυνση των κρατών μελών. Παραδείγματι, η μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης του επεξηγηματικού πρωτοκόλλου στην ε, Σύμβαση της Χάγης ε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα στο ε, portal e e-justice. Κοινή διάσκεψη Επιτροπής και διάσκεψης της Χάγης για το, δημόσιο, για το διεθνές δίκαιο θα, για το δημόσιο διεθνές δίκαιο, συγγνώμη, θα προχωρήσει του χρόνου ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών που ήδη εφαρμόζουν τη σύμβαση που θα μπορέσουν να συζητήσουν τις θέσεις τους και ενθαρρύνεται η κύρωση από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you as well. Uh, any Και εγώ σας ευχαριστώ. Ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Η έκθεση εγκρίνεται. Το Μάρτιο λοιπόν στη Σύνοδο. Now we continue by item 10. Σημείο 10. Ανταλλαγή απόψεων για την προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη και καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακή βία. Το λόγο έχει ο κύριο Μαστάλκα, εισηγητή. <clears throat> pane předsedo, kolegyně το Σεπτέμβριο ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και εκεί με εκπροσώπησε η συναδελφός μου καθώς για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να παρασταθώ πρέπει βεβαίως να κάνουμε το παν για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση αυτή. Αυτή συνεχίζει να είναι η άποψή μου. Είναι η σύμβαση για την πρόληψη της βίας κατά γυναικών και της ανδροκογενειακής βίας που υπογράφει στην Κωνσταντινούπολη το 2011 Πρόκειται για ένα πρώτο ένομο μέσο για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την προστασία γυναικών από όλες τις μορφές της βίας. Και οι στατιστικές στον τομέα αυτό είναι πολύ τραγικές. Το 1 τρίτο των γυναικών, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, γίνεται θύμα 20% έχουν εμπειρίες stalking και διαδικτυακής παρενόχλησης. Τα μέτρα σε αυτόν τον τομέα ανέρχονται σε δύο 228 εκατομμύρια είναι 1,8% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η σύμβαση δεν αναφέρεται μόνο σε γυναίκες, δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Τα συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης εφαρμόζουν το πλαίσιο αυτό και σε παιδιά τα οποία είναι επίσης πολύ ευάλωτα, επίσης σε άνδρες και ηλικιωμένους οι οποίοι επίσης γίνονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι ενδιαφέρον πως μία από τις μελέτες που διάβασα δίνει τα στοιχεία πως 10% των Ευρωπαίων ανδρών παραδέχθηκαν πως έγιναν επίσης θύμα ενδοοικογενειακής βίας, πως είχαν σχετικές εμπειρίες. Σήμερα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή, αλλά την κύρωσαν μόνο 14. Τον Μάιο του 2014 έγινε η πρόταση υπογραφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στο Συμβούλιο δεν προχωρούμε όλοι με τον ίδιο ρυθμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο ενέκρινε μια, ένα κοινό ψήφισμα με το οποίο χαιρετίζει την σκέψη της προσχώρησης στη σύμβαση αυτή. Αυτό είναι όλο. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Συγητή. Ο σκιώδης του SED θα ήθελα να πω μερικές λέξεις γιατί είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση. Η βία κατά γυναικών και η βία λόγω είναι ένα από τα πιο δεδομένα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να θεωρηθεί απειλή για την ασφάλεια της κοινωνίας μας. Έχοντας κατά νου πως το 1 τρίτο όλων των γυναικών στην Ευρώπη είχαν την εμπειρία φυσικής ή σεξουαλικής βίας, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ενηλίκου ζωής τους, και πως 20% των νέων γυναικών ηλικίας 18 έως 29 ετών έχουν βιώσει διαδικτυακή παρενόχληση σεξουαλικού χαρακτήρα, ότι πολλές γυναίκες έγιναν θύματα stalking, μία στις 20 γυναίκες υπέστησαν βιασμό και πάνω από μία στις 10 υπέστησαν σεξουαλική βία. Για να μην αναφερθώ στο ότι πολλά από τα περιστατικά σεξουαλικής βίας δεν αναφερθήκαν καν. Βλέπουμε δηλαδή πως έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνία μας και μάλιστα σε όλα τα κράτη-μέλη αυτά τα φοβερά γεγονότα πρέπει να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου για τους πολιτικούς σε, όλους, σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής, ώστε οι γυναίκες να μην γίνονται πλέον θύματα βίας. Θα ήταν περισσότερο από λάθος εάν εμείς ως πολιτικοί δεν λαμβάναμε αρκετά μέτρα για την πρόληψη του τεράστιου αυτού προβλήματος υπέρ της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν και πιστεύουμε πως είναι κρίσιμη σημασία να επισπεύσουμε την διαδικασία της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας των γυναικών, αντί να σημειωθεί πρόοδος, βλέπουμε μια οπισοχώρηση στην διαδικασία εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Για μένα είναι πολύ ανησυχητικό πως η πολωνική κυβέρνηση του κόμματος της δικαιοσύνη αποχωρεί από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η οποία κυρώθηκε τον Απρίλιο του 2015. Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό μέτρο το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Γι' αυτό και το επίκυρο πολιτικό το οποίο μας λέει πως πρέπει να επισπεύσουμε το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την γνωμοδότησή του χωρίς καμία καθυστέρηση ώστε να ασκήσει περισσότερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση του Κωνσταντινούπολης. Πέραν αυτού πρέπει να θέσουμε προτεραιότητα στα, στα ακόλουθα ζητήματα όπως αυτό αποφασίστηκε στην Ολομέλεια της 24 Νοεμβρίου του 2015 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσω της έγκρισης μιας νομικής πράξης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μπορεί να πρόκειται για μια οδηγία ή για μια άλλη ένομη πράξη, η οποία θα περιέχει ένα σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη σχετικά με όλες τις μορφές βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών και όλης της βίας λόγω ε, χαμηλώντα το, το όριο για την πρόσφαση τη δικαιοσύνη σε αυτό όσο το δυνατόν. Επίση πρέπει να ενεργοποιήσουμε μια ρήτρα μέσω μια ομόφωνη απόφασης η οποία θα ορίζει την βία κατά των γυναικών ως, ε, ως τομέα εγκληματικών πράξεων όπως αυτή ορίζεται στην Συνθήκη της λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει τον λόγο, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. από το τμήμα ισότητας των φύλων και δικαιοσύνης, όπως είπαν οι ομιλητές το ζήτημα είναι σημαντικό που απειλεί την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των γυναικών και υπονομεύει την εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων. Όπως μας λένε οι μελέτες που αναφέρθηκαν μόλις και επίσης ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου το οποίο επιβεβαιώνει το εύρος πολύ προβληματικών προσλήψεων για την διαλογοφύλου σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υπό το πρίσμα μιας εφιστάμενης υγιούς πολιτικής και ενός νομικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου και τρίτον την ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί το ότι οι προεδρίες διευκόλυναν ενεργά τη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις στο Συμβούλιο, γι' αυτό και επικροτούμε την προσέγγιση σχετικά με τη διαδικασία υπογραφή, η οποία αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη βία κατά γυναικών. Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο παράλληλα με την καταπώνηση ενός διοντολογικού κώδικα για την καταπολέμηση της βίας και επίσης για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβαση Επίση, όπω αναφέρθηκε σε προηγούμενε ανταλλαγέ απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν διαφορετικέ πτυχέ όσον αφορά το φαινόμενο. Είμαστε αντιμετωπίζουμε μια σύμβαση η οποία περιλαμβάνει τομεί κοινή αρμοδιότητα αλλά και αποκλειστική αρμοδιότητα είτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για τα κράτη-μέλη. Κυρίω όσον αφορά στον τομέα του ποινικού δικαίου για τα κράτη-μέλη. Η σύμβαση προβλέπει τόσο την προσχώρηση των κρατών μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή η κοινή προσχώρηση δεν χρειάζεται μόνο για νομικούς λόγους, αλλά επίσης για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι να κάνει τη διαφορά για τις γυναίκες στην πράξη. Η σύμβαση αυτή θα γίνει μέρος του, της νομοθεσίας των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Έτσι η φυστάμενη νομοθεσία πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της σύμβασης αυτής. συνάδοντας με την εφαρμογή της οδηγίας περί των δικαιωμάτων των θυμάτων. Επίσης βλέπουμε ένα σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου όσον αφορά τη δυνατότητα δικαιώματος διαμονής παρέχοντας το δικαίωμα σε θύματα να εγκαταλείψουν έναν βίαιο σύντροφο θεωρώντας βία ως ένα στοιχείο ιδιαίτερα δύσκολων περιστάσεων, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να πάρουν μια άδεια διαμονής και να χωρίσουν τον βίαιο σύντροφό τους. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα διαμορφώσει την ερμηνεία. Οι συνέπειες αυτές θα γίνουν σε επίσης στα κράτη-μέλη τα οποία δεν κύρωσαν την σύμβαση. Επί του παρόντος εργαζόμαστε εντατικά για να επιτύχουμε συμφωνία για μια ερμηνεία της σύμβασης με νόημα, η οποία θα καταλήξει στην υπογραφή. Το Κοινοβούλιο ζήτησε την προσχώρηση σε ευρεία, την ευρεία προσχώρηση και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μετά από την το συμπέρασμα σχετικά με την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων θα υπάρξει η αποφασή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση της ε, εφαρμογής της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, μπορείτε να, μιλάτε, να μιλήσετε λίγο πιο σιγά για τους διερμηνείς. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω το αίτημα για ένα ξεχωριστό νομικό εργαλείο με σκοπό την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επί του παρόντος η Επιτροπή θεωρεί πως ήδη υπάρχουν πολλά νομικά και πολιτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του φαινομένου. Αυτή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει επίσης τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η εστίασή μας βρίσκεται τώρα στην εφαρμογή μέτρων που αποφασίστηκαν πρόσφατα όπως η οδηγία περιθυμάτων και η χρήση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως συνεκτικό πλαίσιο για τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της βίας. Η Επιτροπή δεν θεωρεί πως είναι αναγκαίο να προβεί στη θέσπιση περαιτέρω ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό και θα επικεντρώναμε τις προσπάθειές μας περισσότερο στην εφαρμογή της οδηγίας περί θυμάτων και σε άλλους τομείς του ποινικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λεμπρετών, παρακαλώ. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί έχουμε υπερφορτωμένη σε διάταξη και με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα απλώ να επιβεβαιώσω την ανάγκη να καταπολεμήσουμε τη βία εις βάρος των γυναικών. Γιατί είναι πραγματικά ανησυχητικά τα ποσοστά. Μία στις τρεις γυναίκες θα είναι θύμα βία στη διάρκεια της ζωής της. Μία στι τρει και μιλάμε για την Ευρώπη. Φανταστείτε ότι σε άλλε περιοχέ του κόσμου είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Οπότε κάτι οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε. Από αυτήν την άποψη η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη είναι καλό μέσο για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά θα προτιμούσα τα ίδια τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρούν μεμονωμένα στα πλαίσια τη εθνική κυριαρχία στη σύμβαση αυτή και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέλος. Και επίσης ε, υπάρχει ένα ταμπού που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Αυτές οι βιοπραγίες εις βάρος των γυναικών φυσικά γίνονται από άντρε υπηκό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από μετανάστε. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να το πούμε. Φυσικά να καταπολεμήσουμε τη βία ει βάρο των γυναικών, αλλά θα το καταφέρουμε εν μέρει και ε, μειώνοντα δραστικά τη μετανάστευση. Γιατί μεταξύ των μεταναστών ε, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια κουλτούρα που δεν σέβεται τι γυναίκε. Μην ξεχνάμε τι συνέβη στην κολονία και πρόσφατα στο η Γαλλία, όπου μια Γαλλίδα υπήκο υπέστη επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε το θάρρο και το κουράγιο να εντοπίσουμε όλα τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς να παραβλέπουμε κανένα από αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή μας τον κύριο Μαστάλκα, ήθελα να ρωτήσω ε, τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία που μας δώσατε καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ή τα κράτη-μέλη και το Συμβουλίο της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μία έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έγινε το 2014 στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που αφορούν και τις ε, χώρες ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αλλά τα στοιχεία που σας έδωσα εγώ αφορούν τις 28 χώρες μέλη και προέρχονται από το, έρευνα του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωβαρόμετρο. Ο κύριος Μαστάλκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ εν συντομία να σχολιάσω ε, αυτά που μας είπαν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες ε, που θέσαμε και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα οι Επιτροπές ε, Πολιτικών Ελευθεριών και Γυναικών είναι κατ' αρμόδιες, οπότε ε, θα έλεγα να εξετάσουμε στις 21 Μαρτίου και να ψηφίσουμε τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε αυτή την έκθεση στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Ευχαριστώ. Αυτά ως προς την έκθεση του κυρίου Μαστάλκα, τη γνωμοδότηση μάλλον. Και συνεχίζουμε με το σημείο 12, ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης σε σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η συγγετής μας είναι ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή τη για τις εξαίρετες σχέσεις που έχει με τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών πέραν των ε, δηλώσεων των ε, ε, έρωτος με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ξεκάθαρη ότι η εικόνα της, ότι παραγνωρίζονται τα Εθνικά Κοινοβούλια για να μην πω ότι τα βλέπουν αφιψηλού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια απορρέουν άμεσα και νόμιμα έχουν την πιο άμεση νομοποίηση από τον πολίτη αφού εκλέγονται με καθολική ψήφο με ε, καθήκον ε, την επεξεργασία των νόμων και τον έλεγχο της δράσης των κοινοβουλίων ε, στα κράτη τους. Με την αναγνώριση αυτή, αυτής της θεμελιώδους αποστολής εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την αναγνώριση στην αρχή της επικουρικότητας. Πλην όμως, βλέπουμε μια αντίφαση μεταξύ αρχής επικουρικότητας και της αποκλειστικής ε, αρμοδιότητας ε, πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει δράση το ΣΥΠΗΝ, οπότε αυτή το θεωρεί απαραίτητο. Αυτή λοιπόν ε, η παραγνώριση της αξίας και της σημασίας των κοινοβουλίων είναι, είναι οφθαλμοφανής στην έκθεση αυτή το πρόγραμμα εργασίας του 2015 είναι το έγγραφο το οποίο έχουν σχολιάσει περισσότερο τα κοινοβούλια. Δεν είναι αμεληταίο αυτό γιατί το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ε, προγραμματικών δηλώσεων, νομοθετικών προγραμματικών δηλώσεων για όλους μας και τα Εθνικά Κοινοβούλια βεβαίως. Έτσι λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιμένει ότι χρειάζεται βάθος διάλογος πλην όμως ε, δεν αναγνωρίζει την πρώτη στη σημασία της παρουσίας των Εθνικών Κοινοβουλίων, δηλαδή την επεξεργασία του νόμου, αφού δεν τους ε, αναγνωρίζει και θεωρεί ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλία νομοθετικής. Βεβαίω υπάρχουν αντιστάσει από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων και ενδιαφέρον ότι πρόσφατα αυτέ οι εθνικέ αντιστάσει πολλαπλασιάζονται. Ο μηχανισμό επανεγκατάσταση μεταναστών, παραδείγμα που καταγράφεται και στην έκθεση, επευλήθη από την Επιτροπή Juncker, με αποτέλεσμα 12 εθνοσυνελεύσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγυλαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της, Τσέχη, Πολωνή, Σλοβακή και άλλοι ε, μιλούν για παραβίαση επικουρικότητας. Ένα άλλο παράδειγμα του ότι αγνοεί το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν η προσωρινή θέση σε ισχύ τη συμφωνία από πλευρά τη Επιτροπή πριν ακόμη αυτή να κυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πράγμα το οποίο μα συγκλώνησε και νομίζω ότι εν προκειμένου δεν, έγινε, ε, δεν εισακούστηκε η ε, προειδοποίηση τη ε, βουλή τη Βαλωνία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα τελεσίγραφα που επανειλημμένως απευθύνει στην Πολωνία και το Εθνικό τη Κοινοβούλιο η Επιτροπή καλώντας το, καλώντας τη χώρα να ε, κάνει σεβαστές ε, τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται το κράτος δικαίου. Εγώ θεωρώ ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να προβαίνει σταγματικές μεταρρυθμίσεις που θεωρεί σκόπιμες χωρίς να υποχρεούται να κάμπτεται ενώπιον των βουλέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εν τέλει, ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει πάλι πόσο παραγνωρίζει το ρόλο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περίφημη αυτή κραυγή του κ. Γιονκέρ του 2015, περίοδος αναφοράς εν προκειμένου, ε, η κραυγή περί δικτατόρων, που, η δικτάτορα που απευθυνόταν στον κύριο Ορμπάν, δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Όλα αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν πόσο αυθαίρετα συμπεριφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πόσο έχει επιλέξει να υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της τακτικά. Εν όλο, αυτή η αιτήσια έκθεση καταδεικνύει την ε, αλαζονία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπεροψία της έναντι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομολογεί η ίδια το τι πιστεύει για τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί στην έκθεση αυτή τους αναγνωρίζει μόνο ρόλο διασύνδεσης γέφυρας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια για μένα δεν είναι γέφυρες. Είναι ουσιώδη δημοκρατικά όργανα και ως εκ τούτου δεν μπορώ να, εκδώσω, να διατυπώσω θετική γνώμη για την έκθεση αυτή. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σχόλια παρακαλώ από τους συναδέλφους. Ακούσαμε τον εισηγητή. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια. Κοιτάω την κυρία Κάουφμαν. Θέλετε το λόγο. Ναι, πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, πρόεδρε, το σκέφτομαι λίγο πώς θα σας απαντήσω. Γιατί Έχουμε διαφορετικές απόψεις με αυτά που είπε ο κύριος Ντεμπρετών. Τα παραδείγματα που ανέφερε είναι, είναι ανατριχιαστικά όσον αφορά το ΣΕΤΑ. Ξέρουμε, είναι ένα, μια μεικτή συνθήκη. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για το διεθνές εμπόριο. Τώρα, να πούμε, βάσει αυτού του παραδείγματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως δεν σέβεται τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι παράλογο και κανείς δεν θέτει υποπίεση το Πολωνικό Κοινοβούλιο αλλά η Επιτροπή έθεσε, σε έναν μηχανισμό επειδή βλέπει με το δίκιο της έναν κίνδυνο στην Πολωνία, δηλαδή ότι η κυβέρνηση εκεί αμφισβητεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι με αυτή την επιχειρηματολογία αλλά πρέπει επίσης να επιστήσω την, τις πολλές μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ του Κοινοβουλίου μας και των Εθνικών Κοινοβουλίων ότι έχουμε επιτροπές περί Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Εθνικά Κοινοβούλια ότι έχουμε τήσει συναντήσεις διακοινοβουλευτικών επιτροπών και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ διάφορων επιτροπών και πολλά διάφορα άλλα δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη αυτή δηλαδή. Βέβαια, έχουμε πολλά σχόλια από την άποψη αυτή. Δεν ξέρω τι ισχύει στη Γαλλία, αλλά και εγώ εξελέγει σε γενικές εκλογές. Μπορεί ο κύριος Λεμπρετόν να εξελέγει με διαφορετικό τρόπο, όχι δηλαδή σε γενικές εκλογές. Και αυτό το λέω γιατί αρχικά είπε ο κύριος Λεμπρετό ότι είναι καλύτερες οι εκλογές και πιο ε, γενικές για να αναδείξουν τους εθνικούς βουλευτές και δεν ίσχυε το ίδιο για, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ε, και δεν ανακατεύομαι στα εσωτερικά των άλλων χωρών. Αλλά εμεί στη Γαλλία εκλεγόμαστε με βάση ένα πρόγραμμα και ήμουν επικεφαλή του ψηφοδελτίου στην περιφέρειά μου και μάλιστα με εξέλεξαν 500.000 συμπολίτε μου, Γάλλοι συμπολίτε μου. Και με εξέλεξαν για να έρθω εδώ και να αντιταχθώ στο όνομά τους στις απαράδεκτες ε, εξωτερικές ε, παρεμβάσεις στην γαλλική κυριαρχία. Μάλιστα. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 13, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για τις διασυνοριακές αιτήσει επιστροφής έργων και πολιτιστικών αγαθών που λαιλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους. Εγώ πάλι είμαι ο εισηγητής και θα ήθελα να σας πω τα εξής. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών αποφάσισε να δώσει το άδεια στις Επιτροπές ΚΑΛΤ και Γιούρι να συντάξουν νομοθετική έκθεση ε, με αυτό το αντικείμενο. Και δεδομένου του, του περιεχομένου του, του σχέδιου έκθεσης ε, ασχολήθηκα λίγο και με την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση αυτή. Κάποιες πτυχές αυτού του θέματος ε, ίσως εμπίπτουν καλύτερα στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ενιαία αγορά. Άλλες πτυχές του θέματος μπορεί να εδράζονται στο άρθρο 81, παράγραφος 2 της Συνθήκης που αφορά τη συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ε, και διασυνοριακά ζητήματα καθώς και την σύγκληση του δικαίου. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα αυτών των δύο νομικών βάσεων, σε ό,τι αφορά την ακολουθητή διαδικασία. Μια και οι δύο νομικές βάσεις προϋποθέτουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, που με βάση τα πρωτόκολλα 21 και 22 στι συνθήκες ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωρευτικά οι δύο νομικές βάσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα ήθελα να θέσω την ερώτηση στη νομική υπηρεσία μας και να ζητήσω μια γνωμάτευση. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση ασυμβατότητας αυτών των δύο νομικών βάσεων ε, πού θα πρέπει να στηριχτούμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 114 της συνθήκης για του άρθρου ε, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως θα ήταν καλύτερα να προτείνουμε την ε, υιοθέτηση δύο διαφορετικών νομοθετικών πράξεων. Ε, ποιο είναι το προσωρινό χρονοδιάγραμμα τώρα για το θέμα αυτό. Μετά την ε, σημερινή ανταλλαγή απόψεων, και αναμένοντας και την νομική γνωμάτευση για την κατάλληλη νομική βάση τον Απρίλιο. Ίσως η παρουσίαση του σχεδίου έκθεση θα μπορούσε να γίνει στην πρώτη συνεδρίασή μας του Μαΐου, 3 και 4 Μαΐου δηλαδή. Προθεσμοί για τις τροπολογίες 17 ε, Μαΐου, εξέταση των τροπολογιών τον Ιούνιο και ψηφοφορία τον Ιούλιο. Αυτό είναι ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα. Εγώ προτίθεμαι να καλύψω στην έκθεση όχι μόνο προβλήματα του παρελθόντος, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και συναφεί ζητήματα. Θα θέλαμε όμω ε, πέραν του παρελθόντος να προλάβουμε και να επιλύσουμε ενδεχομένω και μελλοντικά προβλήματα από μελλοντικέ δηλαδή συγκρούσει ή ε, ε, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδου λαϊλασίε. ε, υπεξαιρέσεις τέτοιων πολιτιστικών αγαθών να γίνουν στο μέλλον. Γιατί όπως έγινε στο παρελθόν μπορούν κάλλιστα να γίνουν και στο μέλλον τέτοια φαινόμενα, γιατί τέτοιες ε, λαιλασίες πολιτιστικών αγαθών και εργοτέχνης ε, που έγινε στο παρελθόν θα πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθεί και στο μέλλον. Οπότε στο πλαίσιο αυτό ε, σκοπεύω να κάνω μια ανάλυση του φαινομένου αυτού των διασυνοριακών αιτήσεων για επιστροφή αγαθών ε, και να προτείνω κάποιες συστάσεις. Γιατί οι ε, δικαιούχοι, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι κράτη που είναι ε, κάτοχοι αυτών των έργων τέχνης ή να λάβουμε υπόψη τον ειδικό πολιτιστικό χαρακτήρα αυτών των έργων τέχνης. Και τα νομικά ζητήματα αφορούν καταρχήν το εφαρμοστεί δίκαιο που θα πρέπει να ισχύει σε τέτοιου είδου διαφορέ διασυνοριακέ για λαϊλαθέντα αγαθά και να λάβουμε υπόψη και τις, τους περιορισμούς που θα ισχύουν σε τέτοια προβλήματα. Επίσης, οι κανόνες για το βάρος απόδειξης για να αποφασίσουμε κατά πόσο ένα εργοτέχνης ή πολιτιστικό αγαθό έχει γίνει αντικείμενο λαϊλασίας, κλοπής, κατάσχεσης ή παράνομης ε, απόκτησης. Επίσης, τρόπος απόκτησης ε, των σωστών ε, τίτλων ιδιοκτησίας έργων τέχνης ή πολιτιστικών αγαθών και πώς έχουν αποκτηθεί από τους πραγματικούς δικαιούχους. Βέβαια, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι ασύνδετα με άλλες πτυχές του ζητήματος αυτού, γιατί είναι αλληλένδετα και με το προηγούμενο θέμα της λαϊλασίας. Αν αγνοήσουμε λοιπόν μερικές πτυχές δεν θα μπορέσουμε να ε, υιοθετήσουμε μια σφαιρική λύση ε, για το πρόβλημα και το φαινόμενο της λαϊλασίας των έργων Οπότε θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη και τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών που ίσως ε, είναι πιο κατάλληλη για την ανέβρεση δίκαιων γιατί είναι πιο ελαστική και πιο ευπροσάρμοστη στην κάθε περίπτωση και δεν υπόκειται σε ακαμψίες. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να διερευνήσουμε και την δυνατότητα των φιλικών διακανονισμών. Επίσης, δυνατότητα κατάρτισης κοινών συστημάτων, συγκέντρωση στοιχείων για λιλετθέντα, εργατέχνης και πολιτιστικά αγαθά που ενδεχομένως ε, μια τέτοια κοινή καταγραφή διευκολύνει τον εντοπισμό τέτοιων αγαθών και θα διευκολύνει και την παροχή πληροφοριών για την κυριότητα των αγαθών αυτών σε περίπτωση ε, αμφισβήτησης. Αυτά είναι συντομία τα βασικά στοιχεία που θα περιλάβω στην, στην έκθεσή μου, στο σχέδιο έκθεσής μου και περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Και αυτό λοιπόν περιμένω τα σχόλιά σας. Επίσης, ε, θα ήθελα και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας υποστηρίξει και αν ναι, σε ποιες πτυχές πιστεύει ότι θα πρέπει να εστιαστούμε ή για ποια σημεία έχετε διασμούς ή επιφυλάξεις και για ποιου λόγου έχετε τέτοιους ενδιασμούς και επιφυλάξει. Κυρία Γιούτλαντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή του θέματος. Η κυρία Ρωσέρ δεν μπορούσε να είναι παρούσα και έτσι μιλάω εγώ εκ μέρου τη η αποκατάσταση έργων τέχνης ε, ύστερα από λασίες, ε, σε πόλεμες ζώνες είναι μεγάλο πρόβλημα για τις κοινωνίες μας, οι ένοπλες συγκρούσεις ε, διεθνείς είτε εσωτερικές αποτελούν σημαντική απειλή για την πολιτιστική κληρονομιά. Η ιστορία και δυστυχώς και οι σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις έχουν πολλά παραδείγματα να δώσουν για λαιλασία και λαθρεμπόριο κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών, προϊστορικών, ιστορικών, λογοτεχνικών, επιστημονικών. Και αυτό πηγαίνει από την ε, κλοπή, από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς, η μουσεία, ε, καταστροφή, μετατόπιση ε, πολιτιστικών θησαυρών λόγω των πολέμων. Έχουμε πρόσφατα μια άλλη, ένα, μια άλλη διάσταση του προβλήματος, ότι πολλές φορές αυτά τα, τα προϊόντα λαϊλασίας ε, χρησιμοποιούνται και για την χρηματοδότηση των αναπλών συγκρούσεων. Υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν. Η οδηγία 2014-60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών που παράνομα έχουν αφαιρεθεί από την ε, ε, επικράτεια κρατών μελών, αλλά και ο κανονισμός 117.006. Αντίστοιχα, υπάρχουν όμως ζητήματα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, όπως η διεκδίκηση ενώπιση των δικαστηρίων ε, ξένων κρατών, ε, ξένης δικαιοδοσίας, πράγμα το οποίο οφείλεται στο ότι είναι τόσο δύσκολη αυτή η διεκδίκηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει τα νομικά ζητήματα προς την διεκδίκηση μέσω αγωγών για επιστροφή και να προσπαθήσει να δώσει λύσεις ε, δίκες και θεμητές. Η κυρία Ρωσιέ και η ομάδα μας, ε, ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών, προσβλέπει σε πολύ καλή συνεργασία βέβαια με όλους τους συναδέλφους μας για την πολύ σημαντικό το θέμα. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή έχει δήλωση. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Grow. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002-2003 εξέτασε το ψήφισμα που είχε υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν της εκθέσεως Clerk. Ψήφισμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο εξέθεται το πρόβλημα για την αποκατάσταση και διεκδίκηση πολιτιστικών αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εποχή εκείνη είχε επισημάνει πως τα προβλήματα που επεσήμανε η έκθεση αφορούσαν την κυριότητα των έργων τέχνης ή των πολιτιστικών αγαθών ε, και ως τούτου βρισκόταν εκτός του πεδίου εφαρμογής των συνθήκων. Εσείς ε, επισημάνατε στην ομιλία σας ότι τα νομοθετήματα που υπήρχαν να ενισχύει την εποχή αυτή την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν αυτή την εποχή είναι η οδηγία για τα πολιτιστικά αγαθά που ε, αναθεωρήθηκε το Μάιο 2014 με θέση ισχύ τον Δεκέμβριο του 2015. Πλην όμως η οδηγία αυτή αφορά εθνικούς πολιτιστικούς θησαυρού. Αγαθά δηλαδή που ανήκουν σε κράτη. με ιδιαίτερη φύση και καθεστώς ως εκ τούτου. Αν δεν απατώμε, το ερώτημα που εγείρεται με τη νέα σας πρωτοβουλία αφορά πολιτιστικά αγαθά που δεν έχουν το καθεστώς εθνικού θησαυρού. Άρα βγαίνουν από το πλαίσιο εφαρμογή τη οδηγία, Επιπλέον δε αυτή η οδηγία του 2014 60 δεν καλύπτει το ζήτημα τη κυριότητας, το οποίο εναπόκειται στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν. θα σας ε, αναφέρω τον κανονισμό 2015 του 2012 που αφορά τις διαφοράες ως προς τη διεκδίκηση από τον κύριο κλοπημαίων πολιτιστικών αγαθών που προβλέπει αγωγή, πολιτική αγωγή με βάση το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην κυριότητα πολιτιστικών αγαθών και επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να διεκδικήσει την ε, ανάκτηση τέτοιων κλοπημαίων, ε, επιλέγοντας και τη δικαιοδοσία συγκεκριμένα της χώρας στην οποία βρίσκεται το κλοπημαίο αγαθό. Και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα της ε, απαντήσεως της νομικής υπηρεσίας για την αξιολόγηση που τη ζητήθηκε, νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, ώστε να διευκρινιστεί λίγο το ζήτημα της νομικής βάσης που θα επιλεγεί για μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία. Αυτά έχω να πω σε αυτό το στάδιο. Uh, thank you very Ευχαριστώ. Do not see any other... Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο, το 14 τον έλεγχο των κατεξουδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Ο εισηγητής μα είναι ο κύριος Τζαμπάσκι, που απουσιάζει όμως και ζητά συγγνώμη για την απουσία του, θεωρεί πάντως ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουμε σχόλια στην, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εκτελεστικά μέτρα που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού 1382 του 2013 που θεσπίζουν ένα πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη για την περίοδο 2014 με 2020 και τον ε, χρηματοοικονομικό κανονισμό. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Οπότε γίνονται δεκτές οι συστάσεις του εισηγητού μας, του κυρίου Τζαμπάσκη. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 17 τώρα. Ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε μαζί σας τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μια ναι, και έχουμε προβλέψει ότι η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 5 και 4. Ας περιμένουμε καλύτερα ένα-δυο λεπτά ακόμη για να προλάβουν να έρθουν και οι συνάδελφοι που θέλουν να είναι εδώ για την ψηφοφορία. Okay, it's quarter uh, quarter... Είναι πέντε και τέταρτο. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Σημείο 17. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που έχουν την ευθύνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά, γιατί μερικοί ψήφισαν δύο φορές. Και στο υπέρ και στο κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61 τροπολογία που μάλλον έχει απορριφθεί αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές Δεν είμαι βεβαίως για το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Τροπολογία 63. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είδατε που εγκρίθηκε. Ή μάλλον εγώ είδα πως εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 1. Εγκρίνεται, ναι. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 και 87 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 94 άρχεται η ψηφοφορία Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 96. Ποιος είναι υπέρ. Α, Καταπίπτει 96, οπότε πάμε στην 97. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 και 103 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 και 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 108 και 109 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109 9 και 108. 108 και 109 άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τροπολογία 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 και 115 μαζί υπέρ, 113 και 114 συγγνώμη υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται 115 ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 9 δεν είναι αρκετά χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πάλι χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 119 τώρα. Ή μάλλον όχι λάθος. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω χέρια. Να ελέγξουμε την 11. 12 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. Ας επαληθεύσουμε. Ναι. όχι, εγκρίθηκε. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσω. Πιστεύω πως εγκρίθηκε, αλλά σου βεβαιωθούμε. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 133-134 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 135 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 136 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 137 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε παρακαλώ εγκρίθηκε 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ Κατά. Αποχές απερίφθη. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145-146 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 148 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 149 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 150 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 151 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 152-153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 Α, όχι, 152. Ας επαληθεύσουμε. Είχα πει ότι εγκρίθηκε. Ο με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, έχει απορριφθεί. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 155, 156 υπέρ. Κατά. Αποχές αποκλεί, απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 161 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 162 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 163 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 164 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 165 και 166 υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν 21 και 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 175 υπέρ κατά αποχές για να δω νομίζω ότι έχει, ότι έχει κρυθεί αλλά να το επαληθεύσουμε ναι 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αυτό θα το επαληθεύσουμε. Απερίφη. Υπαριθμόν ένα υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά Ας το επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 38 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά το πρώτο τμήμα διορθώνει ο πρόεδρος πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά δεν βλέπω χειρίσκομενο να επαληθεύσουμε

αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ όχι διορθώνω έχει καλυφθεί 50 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το σύνολο του σχεδίου γραμματότης το σύνολό του ηλεκτρονικά Thank you very much. It has been adopted. Ευχαριστώ, εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Χρυσόγωνο. Σημείο 18. Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά επαλήθευση παρακαλώ εγκρίνεται 2 υπέρ συγγνώμη τέσσερα υπέρ τέσσερα επειδή το 2 εκπίπτει εάν εγκριθεί το 3, οπότε γι' αυτό περνάμε στην 4. Ξανά λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 9, υπέρ, κατά αποχές βρισκόμαστε στην εννέα έτσι εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά επαλήθευση παρακαλώ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 αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά συγγνώμη λάθος δικό μου 22 εκπίπτει 20 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Ε, να επαληθεύσουμε παρακαλώ. απορρίφθηκε 25 υπέρ κατά επίσης θα χρειαστεί επαλήθευση εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εντάξει το 27 είπαμε Έχει δίκιο εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι και πάλι είχατε δίκιο εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά επιτρέψτε μου να επαληθεύσω μία φορά ακόμα εγκρίνεται 35 ναι, εγκρίθηκε. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Επιτρέψτε μου να επαληθεύσω και πάλι. Εγκρίνεται και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της όλης γνωμοδότησης εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εαυτό μου Τώρα έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping Τροπολογία 3 υπέρ κατά Να ελέγξω παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μια φορά ακόμα, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης ολόκληρο για τη ηλεκτρονική οδού. Με οριακή πλειοψηφία απορρίφθηκε οπότε ε, δεν μπορώ σε αυτή την περίπτωση να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή Στη συνέχεια έχουμε επιμέρους ψηφοφορίες. Μία το σημείο 20. Για το, για, την, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είναι υπέρ, συγγνώμη, πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Σβιεύκα. 21. Απαιτήσεις για την υποδοχή των ετούμων διεθνή προστασία ηλεκτρονικά. Και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Ζιεύκα εγκρίνεται εντάξει το επόμενο μέρος της συνεδρίασης είναι και κλεισμένο των θυρών οπότε αυτοί που δεν δικαιούνται να βρίσκονται σε συνεδριάσεις και κλεισμένο των θυρών παρακαλούνται ευγενώς να